Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε αυτή τη δημόσια ακρόαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Να καλωσορίσω την Επίτροπο Βέσταγκερ και όλους σας. Και χαίρομαι που αυτή η δημόσια ακρόαση έχει προκαλέσει τόσο ενδιαφέρον. 160 περίπου ενεγράφησαν. Εκπροσωπείται εθνικές αρχές ανταγωνισμού, υπουργεία, ευρωπαϊκές και εθνικές ενώσεις εταιριών, εταιρείες, ομάδες μελέτης, ομάδες συμβούλων. Ένα ιδιαίτερα πολυπληθές και υψηλής ειδίκευσης ε, κοινό για το θέμα μας ε, που είναι η ενίσχυση των εθνικών αρχών ανταγωνισμού για να είναι πιο αποτελεσματικές στην ε, επιβολή της νομοθεσίας. Η πολιτική ανταγωνισμού είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου μας. Στην έκθεση Λάγεν, την ετήσια έκθεσή μας που εγκρίθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι κανόνες που υπάρχουν για τα πρόστιμα για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά, για τα νομικά πρόσωπα πρέπει να συμπληρωθούν και με πρόστιμα για τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται και να είναι αρκετά υψηλά αυτά τα πρόστιμα ώστε να είναι επαρκής ως αποτροπή αυτή η διαδικασία και το Κοινοβούλιο πρέπει να προτείνει τα αναγκαία μέτρα και τονίσαμε ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητες οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού. Θεωρεί ότι αυτό είναι θεμελιώδης σημασίας. Εν ώψη της ακρόασης ε, επίσης ε, παραγγείλαμε και δύο μελέτες για το ρόλο και τις αρμοδιότητες των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού και έχετε και τυπωμένα αντίγραφά τους στην είσοδο της αίθουσας. Και καλωσορίζω και ε, τους ε, υπεύθυνους για τη μελέτη, για τις μελέτες αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δώσει περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες σε αυτές τις εθνικές αρχές για να εφαρμόζουν την πολιτική ανταγωνισμού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εκτιμά ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό αποφασίσαμε να οργανώσουμε μια δημόσια ακρόαση για να συζητήσουμε τα πρώτα αποτελέσματα της ε, διαδικασίας ε, δημόσιας διαβούλευσης που ξεκίνησε η Κομισιόν αρχές του χρόνου. Οι Εθνικέ Αρχέ Ανταγωνισμού είναι εταίροι κλειδί τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή του δικαίου και των κανόνων ανταγωνισμού πριν το 2014 είχαμε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο. Αυτό οδήγησε σε κάποιες δυσλειτουργίες γιατί είχε υπερβολική δουλειά να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από το 2004 και μετά υπήρξε μια μερική αποκέντρωση προς ε, εθνικές αρχές ανταγωνισμού. Τώρα αυτές οι εθνικές αρχές έχουν αναλάβει 85% των αρμοδιοτήτων και λαμβάνω 85% των αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τότε πολλοί θεωρούσαν ότι η αποκέντρωση θα έρθετε εν κινδύνο την ε, ομοιογενή εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το, εθνικό, ε, συγγνώμη, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού. Τώρα είναι γενικά αποδεκτό ότι το δίκτυο μαζί με το αποκεντρωμένο σύστημα λειτουργούν αποτελεσματικά. Αλλά υπάρχουν ακόμη θέματα για το εάν και κατά πόσο οι διαφορές μεταξύ των ε, εθνικών αρχών ανταγωνισμού και των διαδικασιών μπορεί να θέσουν εν κινδύνο τη συνεργασία μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού και την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων. Γιατί ποικίλει πολύ ο βαθμός ανεξαρτησίας, καθώς και το μέγεθός τους, ο προϋπολογισμός τους και το προσωπικό του. Κάποιες είναι ανεξάρτητες και εφαρμόζουν μόνο το δίκαιο ανταγωνισμού, ενώ άλλοι, άλλες τέτοιες αρχές ασχολούνται και με άλλα θέματα, για παράδειγμα προστασία των καταναλωτών και ο βαθμός της ε, ανεξαρτησίας τους ποικίλει. Πολλές εθνικές αρχές ανταγωνισμού δεν έχουν όλες τις εξουσίες που χρειάζονται για να συλλέξουν στοιχεία για παραβάσεις και να οδηγήσουν τη διαδικασία μέχρι τέλους. Δεν μπορούν να βρουν τις εταιρείε που παρανομούν. Επίσης υπάρχουν διαφορές και στα εθνικά προγράμματα επίοικιας που αποθαρρύνουν πολλές εταιρείε από το να παραδεχθούν τις παραβιάσεις αυτές. Θα έχουμε δύο πάνελ κατά τη σημερινή συζήτηση. Η πρώτη ομάδα εργασίας, το πρώτο πάνελ, θα εξετάσει το βαθμό ανεξαρτησίας και τις αρμοδιότητες. Το δεύτερο πάνελ θα εξετάσει τα προγράμματα επίοικιας και τις κυρώσεις στα κράτη-μέλη. Πριν δώσω το λόγο στην Επίτροπο Βέσταγκερ, να σας ε, εξηγήσω και τη διαδικασία για να μπορέσετε να πάρετε το λόγο και επειδή είστε ιδιαίτερα πολύ άριθμοι, θα πρέπει να δείξετε κατανόηση. Δεν θα είναι δυνατόν όλοι να πάρετε το λόγο κατά πάσα πιθανότητα, αλλά θα επιχειρήσουμε να δώσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους το λόγο. Γι' αυτό σας παρακαλώ οι παρεμβάσεις σας ε, να μην υπερβαίνουν τα δύο λεπτά. Φυσικά θα είμαστε ευέλικτοι ανάλογα και το πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσουμε περαιτέρω αυτό το χρόνο ομιλίας. Έχετε πάνω στις θέσεις ε, κάρτες με τις οποίες μπορείτε να μας κάνετε νόημα, αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Οι πορτοκαλιές είναι, συγγνώμη, οι κίτρινες είναι για το πρώτο πάνελ και η ροζ για το δεύτερο θα καθορίσουμε το, τη διαδικασία ως εξής. Θα είναι δύο προσκεκλημένοι μας και μετά ένας ευρωβουλευτής. Υπενθυμίζω ότι η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται ζωντανή στο ίντερνετ και έχουμε διερμηνία σε 20 γλώσσες. Να δώσω το λόγο τώρα στην Επίτροπο Βεστάγκερ για τις αγωγικές της παρατηρήσεις ένα δεκάλεπτο για να μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για την πιο αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού από τι Εθνικέ Αρχέ Ανταγωνισμού. Μάργαρετ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πώ και πώ περίμενα τη σημερινή ακρόαση. σα ευχαριστώ που δείξατε αυτό το ενδιαφέρον και ακριβώ έχετε αφοσιωθεί στο θέμα και ε, έχουμε άλλωστε και τη σχετική έκθεση διότι η Επιτροπή και η Κοινοβούλιο ε, ασχολούμαι με το θέμα, γι' αυτό δείχνει το πόσο σημαντικό είναι. Και οπότε θα πρέπει να δούμε ότι η συνεργασία της Επιτροπής με τις Εθνικές Αρχές ε, είναι μια συμμαχία που είναι πάρα πολύ ισχυρή και είπαμε ότι οι Εθνικές Αρχές λαμβάνουν πολύ περισσότερες αποφάσεις από ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα τα επόμενα βήματα θα είναι πολύ σημαντικά. Έτσι θα εξασφαλίσουμε προς ε, τον κόσμο το να μπορούν να εμπιστευτούν τις ε, αρχές. Οι αρχές να υποπτεύουν την αγορά, να είναι ο ανταγωνισμός ε, και να υπάρχει, υπάρχουν δίκαιοι όροι του παιχνιδιού. Και θεωρώ επομένω ότι είναι όλα αυτά μια πορεία πάρα πολύ επιτυχή και αυτό το οποίο θέλουμε είναι να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε ο πρόεδρος, να δούμε δηλαδή πρώτα-πρώτα το πώς θα καταστεί δυνατόν να έχουν όλε τι εγγυήσει οι εθνικέ αρχέ για να μπορέσουν να, να δράσουν ανεξάρτητα, να έχουν του απαραίτητου ε, πόρου, το προσωπικό, αν έχουν όλα τα εργαλεία που χρειάζεται, ούτω ώστε να πατάξουν ε, κάθε παραβίαση των διατάξεων ανταγωνισμού. Ε, πρέπει να υπάρχει ικανή αποτροπή και να έχουμε κάποια προγράμματα επίοικια τα οποία είναι επίση αποτελεσματικά. Και όλα αυτά μα απασχολούν τόσο διότι δεν θα πρέπει να διαλέγει το που θα εγκατασταθεί σε ποιο κράτος μέλος και αυτό θα αποφευχθεί εάν έχουμε ε, δίκαιους κανόνες ε, στο παιχνίδι του ανταγωνισμού και αυτό αφορά όλες τις αγορές και αυτό και είναι τόσο σημαντικό ε, έχει υποβάλει πολλές ερωτήσεις και σα ευχαριστώ βεβαίω και οι ερωτήσεις σας μας βοηθούν σημαντικά Έχουμε 181 απαντήσεις ε, διαβιβάσει. Αφορούν κάποιες εταιρείες, δημόσιες αρχές, ε, φυσικά πρόσωπα, ε, βιομηχανίες, δικαιωτικά γραφεία και άλλους. Οπότε βλέπετε ότι έχουμε ερωτήσεις από κάθε κατηγορία ενδιαφερομένου για αυτήν την διαβούλευση. Και η γενική μας προσέγγιση έχει πνεύμα πολύ θετικό. Συμφωνία, συμφωνία στη βάση του θέματος ότι δηλαδή θα πρέπει οι εθνικές αρχές να εφαρμόσουν τους κοινωτικούς κανόνες και πάνω από 50% συμφωνούν κατηγορηματικά ή απλώς συμφωνούν ότι θα πρέπει να έχουν αυτό το ρόλο οι εθνικές αρχές. Τώρα, μια άλλη βασική ερώτηση θα είναι το εάν θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Εδώ θέλουμε ένα ισχυρό κίνητρο, γιατί έχουμε πάνω από 75% που συμφωνούν ή συμφωνούν απολύτω, ότι μπορούν να κάνουν περισσότερα οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού. Αυτό αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο, μια σημαντική εφετηρία για την προβληματική μα για το τι μπορούμε να καταφέρουμε. Δύο λόγια τώρα. Για το ποια μέτρα θα βοηθούσαν τις εθνικές αρχές πώς θα μπορούσαν να γίνουν πιο αποτελεσματικές. Πρώτο ερώτημα είναι πάρα πολύ βασικό. Το κατά πόσο θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να έχουμε κάποιες εγγύσεις ώστε να εφαρμόσουμε τις διατάξεις του ανταγωνισμού για προς το συμφέρον της αγοράς του καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά όλα αυτά γίνονται χωρίς να δίνονται οδηγίες προς τούτο πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα. Όπως ξέρετε είναι κάτι το οποίο κάθε τόσο δημιουργεί προστριβές μεταξύ κυβέρνησης και των αρχών των αυτών. Και εμείς λέμε ότι αν δεν έχουμε τέτοιε προστριβέ, πάει να πει αυτό δεν κάνει καλά τη δουλειά, είναι αρκετά αυστηρή η δική αρχή. Και έχουμε, είπαμε, πάνω από 70% που συμφωνούν ή συμφωνούν κατηγορηματικά ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει να και το ευρύτερο θέμα, βέβαια, του πώς λειτουργεί η δημοκρατία. Και αυτό είναι ε, θετικό σημάδι ότι τόσοι πολλοί ε, συμφωνούν στο να υπάρχουν εγγύησεις για ε, την ανεξαρτησία των εθνικών αρχών. Επίση, άλλο θέμα ήταν το πώς θα υπάρχουν ικανοί πόροι για να κάνουν τη δουλειά του αυτέ οι αρχέ. Και 85% των απαντησάντων είπαν ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ικανοί αρκετοί πόροι. Τώρα έχουμε τα εργαλεία, τα εφαρμοστικά και έχουμε πάνω από 85% οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοια μέσα αποτελεσματικά ούτως ώστε να ε, επισημένονται ε, και να διώκονται οι παραβάσεις. Επίσης να υπάρχουν αρμοδιότητες αποτελεσματικές για την επισήμανση των εταιριών που ε, παραβιάζουν το δίκαιο και 80% των απαντησάντων είπαν λοιπόν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και τελευταίο αλλά σημαντικό είναι το θέμα αυτό της επίοικειας. Είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοια αποτελεσματικά προγράμματα και να ενθαρρύνονται οι εταιρείε ε, να αποκαλύπτουν, να, να ε, κάνουν σχετική δήλωση και 85% θεωρούν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ σημαντική αφετηρία, πολύ ισχυρό κίνητρο για μας σε αυτή την προσπάθεια που ξεκινάμε. Τώρα τα αποτελέσματα, οι επιπτώσεις της ε, κοινωτικής νομοθεσίας πάρα πολύ συμφωνούν θα ήταν πάρα πολύ θετικό για την αποτελεσματικότητα, για την εφαρμογή του κοινωτικού δικαίου, τόσο ώστε να υπάρχει ασφαλή δικαίου για τις επιχειρήσεις και επίση να ελαχιστοποιήσουμε τη σχετική δαπάνη, το κόστος για τις ε, επιχειρήσεις και να υπάρχει συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού. Και επομένως οι εθνικές ε, ε, αρχές να βάλουν αποφάσεις οι οποίες να είναι έγκυρες. Οπότε είναι για το θέμα τώρα επενδύσεων και οικονομικής ανάπτυξης και το 80% θεωρεί ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα ωφελήσει ε, επενδύσεις και ανάπτυξη. Βέβαια και άλλα ζητήματα ανέκυψαν ορισμένα, κάθε τόσο ε, αναδύονται και τα γνωρίζουμε από το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ανταγωνισμού και θα πρέπει εδώ να κρατήσουμε το ότι υπάρχει φιλοδοξία να εξισορροπήσουμε από τη μία μεριά την ε, σιδηρά εφαρμογή του νόμου και από την άλλη μεριά να έχουμε δικονομικές ή διαδικαστικές εγγύησεις που και αυτές να είναι α, ισχυρές. Οπότε αυτό το ζήτημα επίση ανακύπτει. Και βέβαια θέλουμε να υπάρχει συνέπεια περισσότερη σε σχέση με το δίκτυο ανταγωνισμού ε, για την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού. Άρα θα πρέπει όλα αυτά να τα λάβουν υπόψη στο μέλλον και αυτή είναι η προσπάθεια εξισορρόπησης. Τώρα, για την πρωτοβουλία αυτή. Τι είδους πρωτοβουλία πρέπει να αναλυφθεί. 64% σχεδόν 65% προτιμούν την αλήψη δράσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εθνικό και μόνο 19% προτιμούν ανάληψη δράσης μόνο από την ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο το 8% θέλουν μόνο εθνικά μέτρα. Πολύ σημαντικό θετικό και αυτό διότι αυτό αναδεικνύει το πόσο έχει κατανοηθεί η σημασία της εργασίας Ένωσης Κρατών και πόσο ακριβώς πρέπει να ενισχυθούν οι κρατικές εθνικές υπηρεσίες. Επομένως, έχει γίνει κατανοητό το τι διακυβεύεται. Και επίσης υπάρχει έντονη επιθυμία ανάληψης δράσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο χρειάζεται οι ελληνικέ αρχές να εφαρμόσουν διατάξεις και ότι αυτά θα πρέπει να προχωρήσουν χέρι-χέρι. Άρα αυτό, αυτό για το μέλλον το έχουμε υπόψη. Και ένα πρόβλημα, μια πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι τότε θα πρέπει να έχουμε ακόμη στενότερη επαφή με τα Υπουργεία των Κρατών Μελών. Μόνο εννέα Υπουργεία μας απήντησαν από κράτη-μέλη. Τα περισσότερα βλέπουν θετικά την προσπάθεια, αλλά θα πρέπει ακόμη να προσπαθήσουμε ούτως ώστε να εμπλακούν και θα πρέπει μέσω του Συμβουλίου να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Και απέδειξε αυτή η διαβούλευση ότι το έργο που επιτελέσαμε μέχρι τώρα είναι αξιόλογο, αλλά και το ότι επιδέχεται βελτίωση. Και όλα αυτά με θετικό πιδοδομικό τρόπο ε, τέθησαν ούτως ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη και τα όσα θα πούμε σήμερα στην ακρόαση. Γι' αυτό και σας λέω ότι αυτή η διαβούλευση υπόσχεται πολλά. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Πράγματι, σας ευχαριστούμε πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σας ως σημειοκίνησης υπόσχονται πολλά και θα περάσουμε στο πρώτο πανέλ ομιλητών. Yes, yes, exactly. So, uh, I know, uh... Ενημερώθηκα ότι η Επίτροπος Φερστάγκερ θα χρειαστεί να αποχωρήσει ε, τώρα και θα δώσω το λόγο στον κύριο Λάιτενμπεργκερ, τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διευθυντής Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Honorable members. Uh, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Σας καλωσορίζω στο πρώτο πανέλ ομιλητών. Στο οποίο θα ασχοληθούμε με τις εξουσίες εκτέλεση των αποφάσεων και την δυνατότητα που έχουν οι αρχές ανταγωνισμού να εφαρμόζουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές ε, ανταγωνισμού, όπως ανέφερε και η Επίτροπος. Πράγματι, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού δεν έχουν πάντα τα εχέγγυα ε, ανεξαρτησίας ή τους απαιτούμενους πόρους για να εφαρμόζουν τις ε, αποφάσεις στα θέματα του ανταγωνισμού. Χρειάζονται λοιπόν αυτά τα δύο στοιχεία και επίσης όλα τα εργαλεία για να καταπολεμούν τις παραβιάσεις από τις ε, επιχειρήσεις στις χώρες τους. Αυτό είναι απαραίτητο για την δίκαιη εκτέλεση των αποφάσεων και την ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε τις ε, απόψεις σας, ποια είναι τα προβλήματα και ποιες λύσεις θεωρείτε ότι είναι βέλτιστες. Θα ξεκινήσουμε την συζήτηση με τους εκλεκτούς μας ομιλητές που εκπροσωπούν τον κόσμο των νομικών, της ε, ε, ενώσεις καταναλωτών, της ενώσεις, ε, τις αρχές ανταγωνισμού και πανεπιστημιακούς. Έχουμε επίσης καλέσει, είχαμε καλέσει έναν εκπρόσωπο του συνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά δυστυχώ ασθένησε και δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί, του ευχόμαστε περαστικά θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Κάνι Φερνάντε, ε, εταίρος στο νομικό γραφείο Κοτρεκάσης Κονσάλες Περέιρα, στο γραφείο Βρυξελών και διευθύντρια για την ομάδα που ασχολείται με τα ζητήματα ε, ευρωπαϊκού δικαίου ε, και ανταγωνισμού. Έχει ε, ιδιαίτερη εμπειρία στα θέματα αυτά. Ε, και ως αντιπρόεδρος ε, της ομάδας αντιτράστ στην, στον Αμερικανικό Δικηγορικό Σύλλογο. Συμμετέχει επίσης και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού. Παλαιότερα έχει υπάρξει και πρόεδρος της Επιτροπής της Ομάδας Εργασίας για τα Αντιμονοπολιακή Νομοθεσία στη Διεθνή Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων. Έχουμε επίσης εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών ως ε, Γενική Διευθύντρια του ΜΠΟΙΚ, λοιπόν, η κυρία Κόιενς, η οποία συμπροεδρεύει στον ε, διάλογο, δι, ε, διατλατικό διάλογο συνεργασία συνεργασίας των ενώσεων καταναλωτών. Μετά, ο καθηγητής Φρεντερικ Ζενή, καθηγητής οικονομικών και διευθυντής της του, του Κέντρου Οικονομικών Μελετών στην σχολή ΕΣΕΚ στο Παρίσι. Παλαιότερα επίσης δικαστής στο Ανώτατο Κυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας. Πρόεδρος επίσης της Ομάδας Εργασίας του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου για το εμπόριο και τον ανταγωνισμό. Έχει ε, επίσης παράσχει συμβουλές σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες σε ζητήματα εμπορικού δικαίου και ανταγωνισμού. Μετά ο κύριος Σαρούνας Κιζεράουσκας, πρόεδρος του Λιθουανικού Συμβουλίου Ανταγωνισμού, με ε, συνεργασία στο παρελθόν ως νομικός σύμβουλος στο ε, Βρετανικό Γραφείο Fair Μετά ο κύριος Μόν, τι καθηγητή της δικαίου ανταγωνισμού ε, στο Ευρωπαϊκό ε, Πανεπιστήμιο στη Φλωρεντία. Επίσης, συνειδητής της ε, ομάδας της Ρώμης για το Ιταλικό δίκαιο, για την Ιταλική αντιμονοπολιακή νομοθεσία. Και τέλος ο κύριος Όλιβε Ρόπκε μάλλον ε, είχε προσκληθεί αλλά δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί. Χαίρομαι λοιπόν που ε, θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τις παρεμβάσεις αυτών των ομιλητών, ο καθένας για έξι λεπτά και δίνω αμέσως το λόγο στην κυρία Κάνη Φερνάντες. Σας ευχαριστώ, η κυρία Φερνάντες. Οι επιχειρήσεις επιθυμούν την σταθερότητα όταν δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου, αυτό δημιουργεί προβλήματα στις επενδύσεις. Όταν έχουμε μια επιχείρηση η οποία λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι δραστηριότητε τη σε κάθε κράτο μέλο θα τύχουν παρόμοια ε, αντίστοιχη μεταχείριση. Αλλά αυτό, αξιολόγηση. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει γιατί οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά τη διαδικασία, όσον αφορά τις αρμοδιότητες τους να εκτελούν αποφάσεις, τις ε, κυρώσεις που επιβάλλουν κτλ. Το οποίο σημαίνει ότι το νομικό πλαίσιο δεν εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο αποτελεί ένα εμπόδιο στην εμπέδωση της ενιαίας αγοράς. έχει αυξηθεί η εναρμόνιση του, ε, της αλλά κατά την άποψή μου αυτό μπορεί να βελτιωθεί. Κάτι το οποίο θα μειώσει όχι μόνο την ανασφάλεια δικαίου και θα βοηθήσει την ανάπτυξη, αλλά θα καθαστήσει και τις διάφορες έρευνες για ε, ε, παράνομες πρακτικές πιο αποτελεσματικές. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού τους απαιτούμενους πόρους για τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση αναθεώρησης του κανονισμού 1 του 2003, θα πρέπει να απαιτηθεί από τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία των εθνικών αρχών ανταγωνισμού και να καθοριστεί ένα ελάχιστο σύνολο αρμοδιοτήτων που θα πρέπει να έχουν οι εθνικέ αρχές ανταγωνισμού. Ε, να αναλάβουν αυτή την υποχρέωση λοιπόν τα κράτη-μέλη. Αυτό θα ενισχύσει και την αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία αυτών των αρχών. Ένας κατάλογος λοιπόν ελάχιστων ε, αρμοδιοτήτων που θα έχουν οι εθνικές αρχές όταν εφαρμόζουν ε, την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον ανταγωνισμό. Έναν ελάχιστο παρανομαστή λοιπόν χρειαζόμαστε. είναι ε, περίεργο, αλλά αυτή τη στιγμή ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών για το πώ ορίζεται η παραβίαση του άρθρου 101-102 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν υπάρχει σχετική εναρμόνιση. Σε ορισμένα κράτη-μέλη, για παράδειγμα, ε, συμπεριλαμβάνονται οι ενώσει επιχειρήσεων, άλλα όχι. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μέλων. Για παράδειγμα, οι αρχές ανταγωνισμού έχουν σε κάτι τη δυνατότητα να ε, διεξάγουν τις έρευνές τους με τεχνικές που δεν είναι αποδεκτές σε άλλα. Επίσης, διαφορές υπάρχουν στις κυρώσεις. Ε, η ίδια ε, πρακτική μιας επιχείρησης μπορεί να τύχει αυστηρής κύρωση σε μια χώρα και να μην τιμωρηθεί καν σε κάποια άλλη οι αρχές, εθνικές αρχές ανταγωνισμού θα πρέπει να ε, προ, ε, οθούν τις ε, πολιτικές, να ζητούν από την κυβέρνηση να εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες να ενισχύουν τον ανταγωνισμό για παράδειγμα ε, εκπονώντας μελέτες ή εκδίδοντας γνωμοδοτήσεις για ε, την αντιμονοπολιακή νομοθεσία ή μια πρόταση τροποποίησης της αντιμονοπολιακής νομοθεσίας, εξολογώντας κατά πόσον αυτή ταιριάζει και με το ευρωπαϊκό πλαίσιο η συνεργασία αυτών των αρχών μέσω του Ευρωπαϊκού ε, Δικτύου Ανταγωνισμού θα πρέπει να γίνεται με τρόπο το οποίο να μην περιορίζει ε, de facto το δικαίωμα ε, υπεράσπισης, τα δικαιώματα υπεράσπισης ε, των επιχειρήσεων. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη εναρμόνιση. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δώσουν τους απαιτούμενους πόρους στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για να μπορούν να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους, όπως περιέγραψα. Το ζήτημα είναι, ο στόχος είναι να καταπολεμήσουμε τα καρτέλ με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε και αποτελεσματικά προγράμματα επί Δεν θα επεκταθώ γιατί θα τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά στο δεύτερο πάνελ. Χρειάζεται, χρειάζονται λοιπόν πόροι και ανεξαρτησία. Εργαλεία και ανεξαρτησία. Το άρθρο 35 του κανονισμού περιγράφει την υποχρέωση των κρατών μελών να ε, στελεχώνουν τις αρχές τους ε, με βάση ε, τα κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό και την αρχή της ισοδυναμίας, έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι αυτές οι προβλέψεις δεν έχουν οδηγήσει σε εναρμόνιση και δεν έχει δώσει τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές να ασκούν τα καθήκοντά τους με αποτελεσματικότητα και χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. Αυτές οι υποχρεώσεις των κρατών μελών ε, θα, θα, θα ήταν περιγραμμένες με τρόπο πολύ πιο ξεκάθαρο από ό,τι είναι περιγραμμένες σήμερα. Θα πρέπει επίσης να αξιολογείται και η απόδοση αυτών των εθνικών αρχών κατά πόσον οδήγησαν οι έρευνές τους σε ποινικέ έρευνες, για παράδειγμα, σε ποινικές διώξεις. Η ευημερία του καταναλωτή έχει αναγνωριστεί ένας από τους κύριους στόχους της πολιτικής ε, ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση λοιπόν ε, του κανονισμού 1 του 2003, πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί και μία αναφορά στην έννοια της ευημερία του καταναλωτή το οποίο θα εξασφαλίσει ότι οι αρχές ανταγωνισμού, οι έρευνες για τυχόν παραβιάσει του ανταγωνισμού δεν θα γίνονται με γνώμονα ε, πολιτικά συμφέροντα ή παρεμβάσει, αλλά με γνώμονα την ευημερία του καταναλωτή. Σα ευχαριστούμε. Κυρία Γκόιν, σας παρακαλώ να τηρείτε τα έξι λεπτά που έχετε στη διάθεσή σα, Ενώ αρχικά είχαμε συμφωνήσει πέντε λεπτά, ήδη έχουμε ένα λεπτό παραπάνω το οποίο μπορέσαμε να σας χορηγήσουμε επειδή δεν ήρθε ο μιλητής από τα συνδικάτα, η κυρία Γκόιενς. Θα κάνω ό,τι μπορώ, λέει η κυρία Γκόιενς. Ευχαριστώ πολύ που καλέσατε την οργάνωση καταναλωτών σε αυτή την ε, ε, ακρόαση. Θα ήθελα να σας πω ορισμένα λόγια για την εφαρμογή της πολιτικής συνταγωνισμού και συμφωνώ με την κυρία Φερνάνδες, σε τελευταία ανάλυση είναι θέμα ε, του κατά πόσο θα ωφεληθεί ο καταναλωτής. Για τον καταναλωτή ο ανταγωνισμός είναι βασικός και τα καρτέλ δημιουργούν προβλήματα. Γι' αυτό οι καταναλωτές χρειάζονται μια ισχυρή πολιτική ανταγωνισμού που να σταματάει τις παραβιάσεις και αν έχει υπάρξει παραβίαση θα πρέπει να υπάρξει και αποζημίωση των καταναλωτών αλλά δεν ε, είναι αυτό το θέμα μας αλλά θα ήθελα να το έχετε υπόψη σας είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της πολιτικής ανταγωνισμού που πολλές φορές παραβλέπεται. Αν δούμε πώς είναι η πραγματικότητα, έχω προετοιμάσει κάποιες διαφάνειες. Αν θέλουμε να δούμε πώς έχουν στην πράξη τα πράγματα, θα διαπιστώσετε ότι δεν εφαρμόζεται σωστά η πολιτική ανταγωνισμού και βλάπτονται οι καταναλωτές αργή η εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού. Θέλει πολύ χρόνο ο εντοπισμός και η επίλυση ενός προβλήματος. Δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι αυτό ισχύει σε όλες τις χώρες. Περισσότερο σε ορισμένες χώρες από άλλες βέβαια. Και είναι κατακαιρματισμένοι οι πόροι. Αν δούμε λοιπόν πώς είναι η κατάσταση των αγορών από την οπτική του καταναλωτή, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλές αρχές που ασχολούνται με τον έλεγχο της συμπεριφοράς στις αγορές. Εμείς εργαζόμαστε με τις αρχές ανταγωνισμού, τις αρχές ε, που ασχολούνται με, τον καταναλω... με τους καταναλωτές, και τις αρμόδιες αρχές για την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, ε, την ιδιωτική σφαίρα. Πολλές φορές υπάρχουν κενά, επικαλύψεις. Και τι διαπιστώνουμε. Οι αρχές αυτές εργάζονται απομονωμένα, δεν συνδυάζουν τις προσπάθειές τους, δεν συντονίζονται για να αξιοποιήσουν καλύτερα τους περιορισμένους πόρους τους. Και υπάρχει διαφορετική εκτίμηση της κατάστασης. Αν υπάρξει κάποια παραβίαση σε ενωσιακό επίπεδο, οι αρχές αντιμετωπίζουν διαφορετικά το πρόβλημα. Και κάτι που θεωρείται παράνομο σε μια χώρα, η προτεραιότητα σε μια χώρα, δεν, δεν ισχύει κάτι τέτοιο σε άλλες. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση τώρα. Δεν θα σας μιλήσω αυστηρά νομικά, παρά το ότι είμαι δικηγόρος, ε, θα επιχειρήσω να είμαι ρεαλιστική. Ένα προφανές ε, μέσο, μια προφανής δυνατότητα που δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς, εδώ και πολλά χρόνια είναι ότι η συνεργασία μπορεί να βοηθήσει για να υπάρξει πιο ενεργή πολιτική ανταγωνισμού. Οι καταναλωτές θεωρούν ότι η συνεργασία των αρχών ανταγωνισμού θα βοηθούσε μέσω της ανταλλαγής ε, συμπερασμάτων και πείρας με τις αρχές ε, για την ιδιωτική σφαίρα, τις τηλεπικοινωνίες, την υγεία. Αυτό ισχύει σε ορισμένες χώρες, αλλά όχι γενικά θεωρούμε ότι δεν είναι μόνο σκόπιμο, αλλά θα γίνει όλο και περισσότερο απαραίτητο. Γιατί αναπτύσσονται οι αγορές, αλλάζουν τα επιχειρηματικά μοντέλα, άρα πρέπει να γνωρίζει πώ έχουν οι ρυθμίσεις για την ιδιωτική σφαίρα όταν προσπαθεί να αντιμετωπίσει μεγάλε εταιρείε ε, τηλεπικοινωνιών, ε, φαρμακευτικέ αν επιχειρήσει, για παράδειγμα, να αντιμετωπίσει αυτέ τι μεγάλε εταιρείε και στον τομέα τη ενέργεια, για παράδειγμα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει περισσότερη ενοποίηση της πολιτικής εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού. Ένα άλλο μέσο που δεν αξιοποιείται αρκετά έχει να κάνει με τη βοήθεια που μπορούν να δώσουν οι οργανώσεις καταναλωτών που γνωρίζουν πολλά για την αγορά. Αυτοί αντιμετωπίζουν ε, τα προβλήματα. Αυτοί έχουν μεγάλη πείρα, ξέρουν πώς μπορεί να καθοριστεί η βλάβη για τον καταναλωτή και έχουν πολλές δυνατότητες να ε, επικοινωνήσουν με πολλούς καταναλωτές και επίσης ε, έχουν και πολύ περισσότερο κύρος έναντι των καταναλωτών σε σχέση με κάποιες δημόσιες αρχές. Πολύ σημαντικό λοιπόν να συνεργαστούμε με τις οργανώσεις προστασίας καταναλωτών, να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας για να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα πενιχρά μέσα μας βλέπουμε ότι στην Ιταλία, την Ολλανδία, τον Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε επιτύχει αποτελέσματα. Γιατί μπορούμε να μην επιχειρήσουμε και αλλού. Αλλά τι διαπιστώνουμε. Ότι υπάρχει απροθυμία εκατέρωθεν και από τις οργανώσεις καταναλωτών και από τις αρχές ανταγωνισμού για να συνεργαστούν. Άρα τι μήνυμα μπορώ να σας δώσω. Επιχειρήστε το να δημιουργήσετε έτσι κλίμα εμπιστοσύνη. ξεκινήστε με άτυπε ε, συνεργασίες σε μικρή κλίμακα για να διαπιστώσετε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε για να βελτιωθεί η εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού σε σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα. Για παράδειγμα, μπορεί να βλέπεστε μια φορά το χρόνο για να καθορίσετε τι προτεραιότητέ σα. Είναι καλό να ξέρουν ε, οι οργανώσει καταναλωτών ποιε είναι οι προτεραιότητε των αρχών ανταγωνισμού. Γιατί τότε και εμεί μπορούμε να αφιερώσουμε προσπάθειε και πόρου σε, αυτές, σε αυτές τις προτεραιότητες των αρχών για να συλλέξουμε στοιχεία και να βοηθήσουμε λοιπόν τις αρχές ανταγωνισμού. Τελευταίο. Η συνεργασία σε ενωσιακό επίπεδο είναι θεμελιώδης γιατί οι διαμεθοριακές ε, παραβιάσεις αυξάνονται συνέχεια. Άρα είναι ουσιώδες να συνεργαστούμε όλοι. Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η δημόσια διαβούλευση για τις αρχές ανταγωνισμού, αλλά ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται και μια επανεξέταση του δικτύου προστασίας των καταναλωτών. Θα ήταν σημαντικό σε αυτήν την αναθεώρηση να επιτύχουμε καλύτερη συνεργασία μεταξύ αρχών ανταγωνισμού και οργανώσεων καταναλωτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο καθηγητής ε, Ζένη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ασχοληθώ με τρία θέματα. Τρία σημεία θα μας απασχολήσουν όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του έργου των εθνικών ανταγωνισμού, η, ανεξαρτησία, οι αρμοδιότητές τους, αλλά και οι πόροι τους. Αλλά αυτά που θα σας πω προέκυψαν από επαφές με ε, πάρα πολλούς παράγοντες του ΩΣΑΠ και δεν ε, συμφώνησαν όλοι αναγκαστικά με τις δικές μου απόψεις. Να δούμε πρώτα πρώτα δύο θέματα μεθοδολογίας τα οποία ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή τι εννοούμε όταν λέμε αποτελεσματικότητα γιατί υπάρχουν ε, ε, πολλές επιμέρους απόψεις, δηλαδή αποτελεσματική χρήση των πόρων, ταχύτητα, διεκπαιρέωσης κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να μην τα ξεχνούμε γιατί προς όλα αυτά τα μέτωπα δεν μπορούμε να κινηθούμε ταυτόχρονα. Άλλο μεθοδολογικό ζήτημα είναι τι εννοούμε για, με το αποτελεσματική αρχή ανταγωνισμού. Τι θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα αποτελεσματικό ή μια υπηρεσία που να είναι πιο αποτελεσματική. Και εδώ δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Ε, ας πούμε, όσον αφορά την διαδικασία, από μια μεριά θα πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών, μπορεί να υπάρχουν ευξημένες δαπάνες, ε, επίσης εκτέλεση αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων και τέλος από θεσμικής πλευράς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την παράδοση της συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Δεν μπορούμε να βρούμε ενιαία λύση για όλους. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε χώρες μεγάλες, χώρες μικρότερες, δεν μπορεί να υπάρξει η ίδια λύση για όλους. Τώρα όσον αφορά την ανεξαρτησία και εδώ θα είμαστε σύντομοι γιατί έχουμε δύο πτυχές της ανεξαρτησίας που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πρώτα-πρώτα όπως αναφέρθηκε η κυβέρνηση, οι κρατικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν ή να επενέσουν ή να αποδοκιμάσουν τις αρχές συνταγωνισμού. Έχουμε το παράδειγμα της ε, Πορτογαλίας όπου κάτι τέτοιο δεν ισχύει αλλά έχουμε και άλλες χώρες όπου η πολιτική αναμεγνύεται στα του ανταγωνισμού. Επίσης θα πρέπει να δούμε κατά πόσον υπάρχει ένα κίνητρο ούτω ώστε αυτοεπαγγέλτος η αρχή του ανταγωνισμού να ασχοληθεί με την ύλη της. Οπότε θα πρέπει να υπάρξουν κανόνες σαφής για την σύγκρουση συμφερόντων. Αλλά επίσης και θα πρέπει να ορίζεται το τι θα απογίνουν τα μέλη μια τέτοια υπηρεσία όταν ολοκληρωθεί η εκεί θητεία του. Τι μπορούν να προσδοκούν κάποια προαγωγή, κάποια θέση, γιατί αυτό βεβαίω και θα επηρεάσει το πώ θα επιτελούν το έργο τους. Στη Γερμανία δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα γιατί στη γερμανική αρχή ανταγωνισμού δεν υπάρχει συνέχεια στην σταδιοδρομία αυτών των υπαλλήλων. Πάντως θα πρέπει και αυτό το θέμα να μας απασχολήσει. Τώρα για να δούμε τις ε, αρμοδιότητες των αρχών αυτών. Θα πρέπει να έχουν μόνο μία αρμοδιότητα, μία λειτουργία ή περισσότερες Εδώ και εδώ έχουμε διαφορετικές λύσεις από κάθε χώρα. Βέβαια και εδώ υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά. Άρα δεν υπάρχει μία και μόνη απάντηση. Τα υπέρ είναι ότι ίσως είναι πιο δόκιμο το να ελέγχει η υπηρεσία αυτή και την ε, ζήτηση αλλά και την προσφορά στην ε, αγορά. Αλλιώς, περισσότερε λειτουργίε έχει περισσότερα μέσα. Και στον ΜΕΟΣΑ έχουν γίνει μελέτες για κάποια θέματα που έχουν προκύψει στον χρηματοπιστωτικό τομέα που πέρασαν από τέτοιες αρχές αλλά δεν έχουν εν στενή ενία σχέση με τον ανταγωνισμό. Και επίση στα μειονεκτήματα ακριβώ ότι όταν έχει πολλέ αρμοδιότητε μια τέτοια αρχή, υπάρχει επιμόλυνση ούτω ή τη μια αρμοδιότητα προ την άλλη. Και άρα δεν θα υπάρξει επάρκεια των πόρων που διαθέσει για να εξυπηρετήσει όλα αυτά τα μέτωπα. Τώρα για να δούμε τι ξέρουμε ε, να λάβουμε υπόψη τι ισχύει και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θα πρέπει και οι αρμοδιότητες να είναι περιχαρακωμένε. Τώρα για να δούμε τώρα τι γίνεται με τους ε, πόρους και την επάρκεια αυτών. Εδώ έχουμε τέσσερα ζητήματα που αναγκυπτουν πρωτα Πρώτα-πρώτα το επίπεδο των ε, οικονομικών πόρων που διαθέσει τη μια τέτοια αρχή ανταγωνισμού και εδώ υπάρχει μεγάλη ποικιλία ανακρατός μέλος. Ούτε αυτό έχει σχέση βέβαια με το μέγεθος της χώρας, αλλά το θέμα είναι κατά πόσον υπάρχει ανεξαρτησία. Δηλαδή, το κατά πόσον η αρχή μπορεί να διαλέξει πού θα κατευθύνει τους πόρους. Υπάρχει και σαν ε, έσοδο βέβαια και η εισπράξη των οικονομικών κυρώσεων, των προστήμων. Για συγχωνεύσεις, ας πούμε, όπως ισχύει σε κάποιες χώρες ή σε Ιταλία και Πορτογαλία. Γιατί αυτό θα δώσει και σταθερότητα στο έργο της υπηρεσίας αυτής. Και ακριβώ ανεξαρτησία σημαίνει το να μπορεί να διαχειριστεί όπως κρίνει σωστότερο του οικονομικού πόρου που έχει στη διάθεσή αυτή. Το εδώ να βάλουμε τελεία, αλλά θέλουμε το εξή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το κοινοβούλιο το τι διαθέτει προ μια τέτοια, ε, τη δεσμεύει τον προπολογισμό για μια τέτοια αρχή ανταγωνισμού, γιατί αυτό πρόκειται να την θωρακίσει και να τη δώσει την σχετική ανεξαρτησία. Και σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Χέσσερα Σα Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχω εργαστεί για δύο ε, αρχές ανταγωνισμού στην καριέρα μου. Η μία ήταν μεγάλη και είχε στη διάθεση τους πολλούς πόρους, η δεύτερη ήταν μικρότερου μεγέθους, επομένω έχω ε, εμπειρία και από αυτά τα δύο σχήματα, μπορώ να σας δώσω μια σχετική παρουσίαση. Η αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων στον τομέα αυτών είναι κάτι το οποίο αφορά και ενδιαφέρει και του εκλεγμένου αντιπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται αποτελεσματικότητα. Έχουμε νέους οι οποίοι ε, εργάζονται πλέον σε αυτές τις αρχές και δεν πρόκειται να συνεχίσουν να επιθυμούν να εργάζονται σε τέτοιου τύπου αρχές εάν δεν βλέπουν ότι η δουλειά τους πιάνει τόπο, δεν έχει αντίκτυπο. Αυτά το θέμα λοιπόν της αποτελεσματικότητας σχετίζεται άμεσα με την ε, ανεξαρτησία και με τους πόρους, με την χρηματοδότηση. Ξεκινώ με το ζήτημα της ανεξαρτησίας. Όταν αναφέρομαι στην αναξαρτησία δεν υπονοώ ότι οι αρχέ ανταγωνισμού λειτουργούν αποκομμένες από την υπόλοιπη κοινωνία. Καθόλου. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν πότε θα δραστηριοποιηθούν, πότε θα αναλάβουν να ερευνήσουν μια υπόθεση χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, χωρίς ε, να δέχονται, ε, να τους υπαγορεύει κάποιος πολιτικός ποια υπόθεση θα αναλάβουν. Επίσης όμως είναι σημαντικό για το ζήτημα της λογοδοσίας. Η λογοδοσία είναι εφικτή μόνο εφόσον η αρχή μπορεί να επιλέγει μόνη της ε, και έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις. Μόνο τότε μπορείτε να αξιολογούνται τα πραγματικά παριστατικά και να λαμβάνετε η απόφαση για το αν θα ερευνηθεί Επίσης, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού, εάν είναι ανεξάρτητες, θα έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην ε, χάραξη πολιτικής για τον ανταγωνισμό. Είναι ξεκάθαρο κοιτώντα την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού δεν ε, είναι εξίσου ανεξάρτητες. Ορισμένες είναι ε, τμήματα Υπουργείων. Άλλες έχουν συσταθεί και λογοδετούν στην κυβέρνηση και άλλες είναι εντελώς ανεξάρτητες αρχές. Ένα στοιχείο είναι όμως η ανεξαρτησία στο νομικό πλαίσιο και ε, άλλο στοιχείο είναι, άλλο θέμα είναι εάν επί του ουσίας de facto είναι ανεξάρτητη η αρχή. Την πραγματική ανεξαρτησία είναι αυτή που θα πρέπει να επιδιώκουμε. Και αυτό εξαρτάται από την πολιτική νοοτροπία στις, στην κάθε χώρα οι οποίες νοοτροπίες διαφέρουν κατά πολύ όπως γνωρίζετε. Θα σας παρουσιάσω την εμπειρία μου από τη Λιθουανία. Στη Λιθουανία δεν είναι σπάνιο ένας πολιτικός να σχολιάσει δημοσίως τις ε, επιλογές μιας αρχής όπως η δικιά μας, το γεγονό ότι ανέλαβε ή όχι να διερευνήσει μια υπόθεση. Δεν υπονοώ ότι η ανεξαρτησία στον νόμο δεν έχει σημασία, Αντιθέτω, εάν υπάρχει ανεξαρτησία κατοχυρωμένη νομικά, αυτό μας δίνει ένα βήμα, ένα εργαλείο στο οποίο μπορούμε να αναφερθούμε, μπορούμε να το επικαλεστούμε αν χρειαστεί. Και η νομικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία θα πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο διατυπωμένη ώστε να μην μπορεί ένας πολιτικός να παρακάμψει τις διατάξεις του νόμου. Οι αρχές ανταγωνισμού προσπαθούν να καταπολεμήσουν τον περιορισμό του ανταγωνισμού και αυτό συμπεριλαμβάνει όμως και πολιτικές που λαμβάνει η ίδια η κυβέρνηση, οι δημόσιες πολιτικές για τον περιορισμό του ανταγωνισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να παρεμβαίνει η αρχή. Όσον αφορά τους χρηματικούς πόρους, είναι σημαντικό ο προϋπολογισμός της ε, αρχής να είναι ανεξάρτητος από ε, την της κυβέρνησης, αλλά και αυτό δεν αρκεί. Χρειάζονται κανόνες πιο εξειδικευμένοι. Για παράδειγμα, οι οποίοι δεν θα επιτρέπουν σε μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι, έχει δυσαρεστηθεί από την πρωτοβουλία που ανέλαβε μια εθνική αρχή ανταγωνισμού να τις επιβάλλει αντίπεινα, να τις περιορίσει τη χρηματοδότηση αφενός και αφετέρου χρειαζόμαστε κανόνες για την αυτόνομη και αποτελεσματική χρήση των πόρων που είναι στη διέθεση των ε, αρχών. Πολύ συχνά οι εθνικές αρχέ ανταγωνισμού δεν έχουν τους απαιτούμενους χρηματικούς πόρους, ούτε για ε, μισθούς, είτε για χώρους, είτε για να διεξαγάγουν έρευνες. Συμπερασματικά, για να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή των κανόνων για τον ανταγωνισμό. Χρειάζεται ανεξαρτησία στο νομικό πλαίσιο, αλλά και στην πράξη. Και αυτό είναι μια διαδικασία συνεχής, διαρκής. Δεύτερον, οι αρχές ανταγωνισμού θα πρέπει να έχουν πόρους στη διάθεσή τους με τρόπο προβλέψιμο και ανεξάρτητο. Και τέλος, η ανεξαρτησία και η επαρκή χρηματοδότηση των αρχών θα πρέπει να συνδυάζεται με επαρκή λογοδοσία. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον καθηγητή Μόντι, τελευταίο ομιλητή σε αυτό το γύρο, σας υπενθυμίζω ότι μετά του ομιλητέ μας θα έχετε εσείς το λόγο για να κάνετε παρεμβάσεις, ερωτήσεις, για να δηλώσετε ότι θέλετε το λόγο. Παρακαλώ συμπληρώστε μία κάρτα ομιλίας για να σας καλέσουμε να πάρετε το λόγο την κατάλληλη στιγμή. Παρακαλώ, ε, καθηγητά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την δυνατότητα συμμετοχής για να βοηθήσω την προσπάθεια να εφαρμοστεί ο νόμος. Ε, πρώτα απ' όλα θέλω να μιλήσω για τις επιπτώσεις που είχε στην, ε, ο κανονισμός 2001 στην εφαρμογή του νόμου. Νομίζω ότι υπερβάλλουμε τον τρόπο με τον οποίο ε, έχουν γίνει αυτές οι προσπάθειες. Αν εξετάσουμε πιο στενά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν οι εθνικές ε, αρχές ανταγωνισμού πριν και μετά τον κανονισμό 1-2003, θα διαπιστώσουμε ότι ακόμη και πριν την εφαρμογή του κανονισμού ήταν ενεργές οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού για να εφαρμόζουν το δίκαιο ανταγωνισμού στις χώρες. Αν μελετήσουμε προσεκτικά την ε, δουλειά αυτών των αρχών, προκύπτει ότι ακόμη και πριν αλλά και μετά το 2004 ασχολούνται με τοπικά καρτέλ και τοπικές συμφωνίες ε, διανομής. Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή από τις εθνικές αρχές ασχολεί, ασχολείται με τις εθνικές αγορές. Η εφαρμογή του ενωσιακού νόμου παράλληλα δεν είχε αποτέλεσμα επί της ουσίας, ούτε επί των προστήμων των εθνικών αρχών και σε κάποιες δικαιοδοσίες, περίπου μισές, αν όχι παραπάνω από τις αποφάσεις των εθνικών αρχών, βασίζονται μόνο σε εθνικό δίκαιο γιατί οι παραβιάσεις δεν είχαν επιπτώσει σε ενωσιακό επίπεδο, οπότε δεν ισχύει ο ενωσιακός νόμος. Τι σημαίνουν όλα αυτά τώρα για οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία. Πρώτα είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι οι εθνικέ αρχέ βοηθούν για να βοηθήσουν πιο ανταγωνιστικέ ευρωπαϊκές αγορέ ακόμη και πριν τον εξυγχρονισμό. Η δραστηριότητα αυτών των αρχών υποτιμάται αν υπολογίζουμε μόνο τις περιπτώσεις όταν εφαρμόζουν ενωσιακό νόμο, γιατί η εφαρμογή του εθνικού δικαίου ανταγωνισμού κάνει την ευρωπαϊκή αγορά πιο ανταγωνιστική. Δεύτερον, αν θέλουμε μια νέα οδηγία που θα δώσει νέε αρμοδιότητε στι ελληνικέ αρχέ για να εφαρμόσουν τον ενωσιακό νόμο ανταγωνισμού, θα έχουμε μια νέα συμμετρία. Δηλαδή θα έχουν διαφορετικέ αρχέ, ανάλογα, διαφορετικέ αρμοδιότητε, καλύτερα, ανάλογα με το αν εφαρμόζουν εθνικό ή ενωσιακό νόμο. Δηλαδή, οι αρχές που εφαρμόζουν ε, κυρίως ε, εθνικό δίκαιο, δεν θα επηρεαστούν καθόλου από ένα νέο νοσιακό νομοθέτημα. Άρα αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Οι εθνικές αρχές χρειάζεται να εφαρμόζουν μόνο τον ενωσιακό νόμο, μόνο όταν υπάρχουν ε, ενέργειες διενωσιακές. Κάτι άλλο. Όλες περίπου οι εθνικές αρχές εκτός από μία μπορούν να εφαρμόσουν ε, πρόστιμα μόνο για πολιτικές κατά του ανταγωνισμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι μόνο εάν υπάρχουν ενουσιακές παραβιάσεις μπορούν να εφαρμόσουν ε, ε κυρώσεις. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του ε, καρτέλ αλευριού. Δεν θα ήταν καλύτερα να υπάρχει μία εθνική αρχή ανταγωνισμού που να ορίζεται ως η αρμόδια για να εφαρμόσει τον ενωσιακό νόμο εφόσον υπάρχουν διαμεθοριακές επιπτώσεις. Αυτή η δυνατότητα για να μπορούν να εφαρμόζουν οι εθνικές αρχές και έξω εδαφικά τον ουσιακό νόμο, θα ενίσχυε το ρόλο τους. Δεύτερο σχόλιο. Μέχρι τώρα η συζήτηση ασχολείται με τις δυνατότητες ε, να εφαρμόζουν κυρώσεις οι αρχές αυτές. Μία άλλη δυνατότητα που θα μπορούσαν να έχουν θα ήταν να κάνουν αποφάσεις για μη παραβίαση. Πολύ συχνά μία έρευνα αποκαλύπτει ότι κάποια συμφωνία ή κάποια πρακτική δεν είναι κατά των διατάξεων. Όπως έχει τώρα ο νόμος, οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να λάβουν μια θετική απόφαση, να πούν όχι, δεν υπάρχει παραβίαση. Θα μπορούσαμε να αναθεωρήσουμε τον κανονισμό 1-2003 για να δώσουμε αρμοδιότητες στις εθνικές αρχές να λαμβάνουν και τέτοιες θετικές αποφάσεις. Τρίτο σχόλιο. Πώς ε, να βελτιστοποιήσουμε τη συνεργασία μεταξύ αυτών των εθνικών αρχών. Όπως ακούσατε, το δίκτυο των αρχών ανταγωνισμού ενίσχυσε το κλίμα εμπιστοσύνη και δημιούργησε δυνατότητε επικοινωνία. Αλλά το δίκτυο δεν έχει επαρκή ε, λογοδοσία. Αλλά το βασικό είναι πώ να ενισχύσουμε την ε, συνεργασία και τον συντονισμό. Για παράδειγμα, πρόσφατα τρει εθνικέ αρχέ εξέτασαν ορισμένε επιγραμμικέ πλατφόρμες κρατήσεων. Τρει αρχέ έλαβαν τρεις ε, διαφορετικές αλλά ταυτόσιμες αποφάσεις συμβασμού οι οποίες έγιναν δεκτές από όλες εκτός από μία από όλες τις άλλες αρχές ε, ανταγωνισμού σε εθνικό επίπεδο. Άρα η συνεργασία και ο συντονισμός είναι η καλύτερη λύση μέχρι στιγμής ή λόγω των περιορισμένων πόρων της Κομισιόν και των εθνικών αρχών θα ήταν καλύτερα μία εθνική αρχή να επιφορτιστεί με την εξέβρεση λύσης που να ισχύει για όλους. Και δεύτερον, Πρέπει όλε οι εθνικέ αρχέ να συμφωνούν για το πώ ε, να ρυθμίσουν μια περιοριστική πρακτική. Βέβαια η ασφάλεια δικαίου θα έλεγε ε, βεβαίω πρέπει. Αλλά η εμπειρία για το πώς ο καθένα μπορεί να λύσει το πρόβλημά του μπορεί να βοηθήσει. Αυτέ είναι οι δύο ερωτήσει που ίσω θέλατε να εξετάσετε. Για να δούμε πώ μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε το παρόν σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τα πέντε μέλη του πάνελ για όσα ενδιαφέροντα μας είπαν που σίγουρα εμπνέουν προς συζήτηση. Ο πρόεδρος μας είπε ότι θέλουμε να λάβουν το λόγο και ευρωβουλευτές και άλλοι προσκεκλημένοι μας. Πάντως προς το παρόν η συντηρητική πλειοψηφία των εχόντων ζητήσει το λόγο είναι ευρωβουλευτές. Σας υπενθυμίζω πάντως ότι μπορεί να ζητήσετε τον ε, λόγο συμπληρώνοντας αυτό το δελτίο, αυτή την έγχρωμη καρτούλα. Πρώτος, έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος ε, Μάιερ και έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ θέλω να αναφέρω τρεις παρατηρήσει και μία ερώτηση πρώτα-πρώτα όσον αφορά την ανεξαρτησία. Ανεξαρτησία τι είπα να πει. Πρώτα-πρώτα θεσμική ανεξαρτησία και από την άλλη μεριά υπάρχει και η προσωπική ανεξαρτησία. Πολύ σημαντικά και τα δύο. Το πρώτο μπορεί να περιχαραγωθεί από τον νόμο, το δεύτερο όμως δύσκολο να επιτευχθεί. Επίση, υπάρχει γίνεται ε, προσπάθεια να έχουμε μια μεριά την λογοδοσία, μια μεριά την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, αλλά θα πρέπει επίση να θυμόμαστε γιατί χρειάζεται η βιομηχανία και οι εταιρείε, χρειάζεται να υπάρχει προβλεψιμότητα, άρα χρειάζεται να υπάρχει κάποιο ε, διάστημα ε, χρονικό στο οποίο να δεσμεύεται η υπηρεσία θα εκδώσει απόφαση. Επίση κάτι άλλο που αφορά τον, τον ανταγωνισμό, την ε, ελεύθερη οικονομία, που ε, και αυτά βέβαια είναι βασικά για μας, γιατί υπάρχουν στην Ευρώπη πάρα πολλοί απαγορευτικοί κανόνες δικαίου που ε, πνίγουν την ε, αγορά και οδηγούν στην συζητηθήσα κατάτμιση, ας πούμε, στους σειροδρόμους ή στα ενεργειακά, πολύ σημαντικά. Τώρα, έχω μια ερώτηση. Άμα δω την έκθεση, την την περσινή, βλέπουμε τι λέει για την ψηφιακή οικονομία, την ενέργεια και την ε, φορολόγηση. Εκεί στάθηκα. Γιατί θα πρέπει να δούμε ε, ότι τελικά εξορισμού υπάρχει προστιβή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις Εθνικές Αρχές ή με την ε, κυβέρνηση. Γιατί υπάρχει αυτό το πάγιο πρόβλημα του τι φορολογική πολιτική ακολουθεί κάθε κυβέρνηση. Άρα και εκεί θα πρέπει να αναπτύξουμε κάποια δραστηριότητα και να φροντίσουμε να υπάρχει αποτελεσματικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βουλευτά. Ο επόμενο που έχει δει τον λόγο, ο κύριο Αλφρέντ Τσάντα. Ευχαριστώ. Ερώτηση. Ήρθε στην ώρα της αυτή η συζήτηση. Από πολιτικής πλευράς όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε κεντροκατευθυνόμενη πολιτική ανταγωνισμού και εναρμόνιση όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση των σχετικών διατάξεων. Όμως, λέει ο κύριο Σάντ, είναι λεπτή η κατάσταση. Είδατε τι προέκυψε ε, στην Ευρώπη όσον αφορά τις σχέσεις ε, κρατών και Βρυξελών σε σχέση με αρμοδιότητες, δικαιώματα, κάστο. Άρα, είδατε πώς μπορεί να ερμηνευτεί η πρωτοβουλία αυτή τώρα. Τώρα κάτι άλλο, όσον αφορά τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού σε σχέση με την γραφειοκρατία των Βρυξελών που λέμε. Μπορούμε να πετύχουμε μια εξισορρόπηση. Βελικά, το πώς κανείς διαμορφώνει πολιτική ανταγωνισμού ε, θα καθορίσει κατά πόσον θα έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι η ίδια αρχή. Κάτι άλλο τώρα που αναφέρθηκε. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το τι ισχύει όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις. Φυσικά και δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να υπάρξει ενιαία προσέγγιση για όλα τα κράτη. Όμως λέμε τώρα για μια νέα προσέγγιση όσον αφορά τις εθνικές φορολογικές πολιτικές. Και όλα αυτά είναι άξονε άξονες πάνω στους οποίους κινείται η γραφειοκρατία των Βρυξελών. Άρα, αυτό θα πρέπει να προσέξουμε τώρα και όχι να προχωρήσουμε μπροστά για νέες προβλέψεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βουλευτάλη, ο Πρόεδρος. Ο επόμενος. Έχετε το λόγο. Είναι κύριο Λόγκη από το, κύριο, από το ECR. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση που σχετίζεται με την ανεξαρτησία των αρχών ανταγωνισμού. Θέλω ιδιαίτερα να ασχοληθώ με το θέμα της ε, ανεξαρτησίας του προϋπολογισμού τους. Δηλαδή πόσους πόρους έχουν στη διάθεσή τους αλλά και τι στα σταδιοδρομίας έχουν ε, αυτοί που εργάζονται σε αυτές τις υπηρεσίες, ανάλογα με το τι αποφάσεις παίρνουν. Με ενδιαφέρει αυτό, διότι αυτός που καθορίζει τον προπολογισμό αυτών των ε, αρχών, πολλές φορές είναι κατηγορούμενος. Για παράδειγμα, για τις ανανεώσιμες ενέργειες στην Γερμανία. Τίθενται διάφορα θέματα, τρομερά πολιτικής ανταγωνισμού που έχουν φτάσει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και κατά τη γνώμη μου οι αποφάσεις που λήφθηκαν δεν είναι ικανοποιητικές, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι σαφές ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ε, το κράτος είναι και δικαστής και κατηγορούμενος. Γι' αυτό θα έπρεπε να σκεφτούμε κάποιες καινοτόμες μορφές χρηματοδότησης των αρχών ανταγωνισμού. Θα ήθελα, επειδή υπόθηκε αυτό σε κάποιο κείμενο, να μου πείτε τι ακριβώς εννοείτε. Για παράδειγμα, θα μπορούσα να σκεφτώ ότι θα μπορούσε να καθορίζεται ένα ποσό από το διακύβευμα που να χρηματοδοτεί ακριβώς ε, τους οργανισμούς. το ύψος αυτής της συμμετοχής ε, θα μπορούσε να καθορίζεται από έναν εξάρτητο οργανισμό με αντικειμενικά κριτήρια. Αυτό θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον κρατικό προπολογισμό, την κρατική χρηματοδότηση. Έτσι θα μπορούσε να υπάρξει μια αποδέσμευση των αρχών αυτών από τις πολιτικές πιέσεις. και από το γεγονός ότι παίζει ρόλο ε, για την ε, πολιτική ανταγωνισμού τελικά το ίδιο το κράτος. Ε, άρα εμπλέκεται. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Βεν Γκίγκολτ, Τον Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα σε σχέση με την ανεξαρτησία το απευθύνω σε όλους τους ομιλητές. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την ε, ανεξαρτησία στον τομέα του ανταγωνισμού. Όταν υπάρχουν ιδιωτικοποίησεις, όταν από ένα δημόσιο, μη δημόσια υπηρεσία ε, μεταβαίνουμε στον ιδιωτικό τομέα. Όταν κάποιο υπάλληλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή φεύγει από την Επιτροπή και ε, εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, δεν έχει τη δυνατότητα φυσικά να ασχοληθεί με την ίδια υπόθεση με την οποία ασχολείται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά μπορεί πάντα να συνεχίσει να ασχολείται με παρόμοιε υποθέσει και έχουν υπάρξει τέτοια περιστατικά, όπου προφανώ υπάρχει ε, σύγκρουση συμφερόντων. Προφανή. Θα ήθελα λοιπόν την άποψή σας για το πώς ε, έχει αυτό αντιμετωπιστεί στα διάφορα εθνικές δικαιοδοσίες, ε, στα κράτη-μέλη, εάν έχουν βρεθεί καλύτερες λύσεις και ποιες είναι οι προτάσεις σας, οι στάσεις, τι θα έπρεπε να γίνει. Ευχαριστούμε τον ε, αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου. Μετά από αυτές τις παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών έχουν ζητήσει δύο συμμετέχοντες το λόγο. Πρώτα ο κύριος Τίσενπλομ ε, από την Σουηδική Αρχή Ανταγωνισμού. Please use the... Μπορείτε παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο. Thank you. Now you hear me. Με ακούτε τώρα. Σας ευχαριστώ. Πρώτα πολύ να συγχαρώ την ε, Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για τη διοργάνωση αυτή τη πολύ σημαντική συνάντηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμετοχή τη. Πιστεύω ότι τα άρθρα 101 και 102 τη ε, συνθήκη είναι πολύ σημαντικά για την εμπέδωση τη ενιαία αγορά στην Ευρώπη, ε, η οποία παρέχει μια σειρά επιχειρηματών στου πολίτε τη Ευρώπη, ευημερία κτλ. Προσωπικά έχω εμπειρία, ε, μιας και έχω εργαστεί επί έξι χρόνια ε, στη παλαιότερα είχα εργαστεί στην ε, Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής και τώρα εδώ και έξι χρόνια εργάζομαι στην Σουηδική Αρχή Ανταγωνισμού. Τα θέματα λοιπόν που συζητούμε σήμερα με έχουν απασχολήσει, το δυνατότητα που έχουν οι αρχές ανταγωνισμού να διεξάγουν έρευνες, η ανεξαρτησία τους, οι πόροι τους, η ανεξαρτησία από οποιαδήποτε παρέμβαση η οποία ε, δεν είναι αποδεκτή. Και εν τέλει είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές μεταξύ των συστημάτων σε κάθε κράτος μέλος. Είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε αυτό στους Ευρωπαίους πολίτες. Γιατί τελικά κάποιους πολίτες σε κάποια χώρα να υποφελείται από έναν υγιή ανταγωνισμό και άλλοι αλλού να μην το έχουν αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι σήμερα μπορούμε να ξεκινήσουμε ε, μια, ενδιαφέροντα διάλογο. Έχουν μια ευκαιρία να το πράξουν αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε τελικά αυτές οι θεμελιώδεις αρχές να επωφελήσουν όλους τους πολίτες σε ολόκληρη την Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριος Χωσερίβας. Έχετε δύο λεπτά. Παρακαλώ με το μικρόφωνο. Μιλήστε. Είναι το κουμπάκι στα δεξιά, όπως βλέπετε το μικρόφωνο. Πρέπει αυτό να πατήσετε. Α, αυτό είναι. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση. Αφορά κάτι που ο καθηγητής Ζενή ανέπτυξε τότε που είπε ότι το ερώτημα είναι τι αναζητούμε πιο αποτελεσματικό σύστημα ή πιο αποτελεσματική υπηρεσία ή αρχή, γιατί αυτά δεν ταυτίζονται. Και μια που έχω κάνει μαχόμενη δικηγορία, εγώ θα ήθελα ε, την πρώτη εκδοχή, ένα αποτελεσματικό σύστημα. Δεύτερη το ερώτηση που έχει σχέση με τις ε, σχετικές διαδικασίες γιατί διάφοροι από το πάνελ ανέφεραν στο ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ της κάθε χώρας όσον αφορά τη διαδικασία, τις παρεχόμενες εγγυήσεις. Οπότε το ερώτημα που αναδύεται είναι κατά πόσον τα δικονομικά δικαιώματα των ε, εταιριών ε, για το δίκαιο ανταγωνισμού είναι δικαιώματα τα οποία είναι δικαιώματα για τα οποία υπάρχουν εγγύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης θέλω να πω ότι δεν είχαμε στην διαδικασία σε πάρα πολλά κράτη-μέλη ε, πρόβλεψη για ένσταση από πλευρά της ε, εταιρεία. Τελικά με την ε, πρακτική των δικαιωτικών δικαστηρίων άλλαξε η κατάσταση σε συγκεκριμένο κράτος μέλος Τώρα όμως αυτό καταργεί. Τώρα δεν ξέρω εάν υπάρχει τελικά στην συγκεκριμένη χώρα ε, αυτού του είδους ε, η δήλωση ένστασης. Επόμενος θα πρέπει να έχουμε και εξεγγυήσεις για τα δικαιώματα των διαδίκων, θα πρέπει να υπάρχει κάποια διαδικασία για ε, αίτηση πληροφοριών. Έχουμε το θέμα της ε, εγγράφου ή προφορικής απαντήσεως, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Δεν θα πρέπει οι εθνικές αρχές επίσης να, να διέπονται από ένα σύστημα εγγύσεων σε σχέση με όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και κατόπιν όσον ακούσαμε από το ακροατήριο ξαναγυρίζουμε στο, ε, στους, ε, ευρωβουλευτές και έχεις δει στο λόγο ο κ. από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε. Και όλοι οι ομιλητές μας είπαν ότι χρημάτων και πόροι γενικότερα και ο κύριος Ζενή μας είπε ότι δεν μπορούμε να έχουμε ενιαία λύση για όλους. Οπότε και εγώ τώρα προβληματίζομαι για μια χώρα όπως η, ε, μια χώρα όπως η, η Ιρλανδία που είμαστε 4-5-6 εκατομμύρια. Τι, τι θα, θα έχουμε δύο αστυνομικού που αρκούν για όλη τη χώρα σύμφωνοι, δεν υπάρχει ενιαία λύση, αλλά αρκεί κάτι τέτοιο για μας, γιατί προβληματιζόμαστε πολύ στη χώρα μας για το πώς θα εφαρμοστεί το δίκαιο του ανταγωνισμού. Γιατί ξέρετε από το 2005 ο σημερινό επιτροπής ο κύριο Χογκάν είπε ότι υπάρχει πρόβλημα με το δίκαιο ανταγωνισμού μας. Το είπε στο κοινοβουλίο μα. Και θα πρέπει αυτό να το ξανακοιτάξει κανεί. Αυτό για την αγόρευση του νευρίου του 2005. Να το ξανακοιτάξει ο κ. Σόγκαν διότι δεν άλλαξε η κατάσταση. Δεν υπάρχει υπηρεσία για εφαρμογή του δικαίου. Ε, ε, μας 24 δις από τότε. Αυτή η μη εφαρμογή. 4,5 εκατομμύρια είμαστε και έχουμε μόνο δύο ε, αξιωματικού, μόνο δύο υπαλλήλους για ε, στις υποθέσει ανταγωνισμού. Και αυτοί που έχουν ζημιωθεί από τα καρτέλ παλεύουν να αλλάξει ο νόμος. Κάποιος είχε προσπαθήσει να προσφύγει και στα δικαστήρια. Επί 20 έτη έδινε δικαστικό αγώνα, αλλά ήταν ε, τέτοιο το βάρος ε, της αποδείξεως γιατί τελικά έγινε ποινικό το δικαστήριο που δεν έβγαλε άκρη. Καταλαβαίνω ότι αυτό γίνεται στα πολιτικά δικαστήρια στα περισσότερα κράτη-μέλη. Άρα, μήπως κάποιο από το πάνελ να μας πει τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει στην Ιρλανδία. Είναι δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι στη χώρα μου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βουλευτά. Εδώ ολοκληρώνουμε τις ερωτήσεις και να δούμε μήπω κάποιο άλλο θα ήθελε από το κρατήριο να λάβει το λόγο. Α, να. Βλέπω τον κύριο Σουβάμπ του Λαϊκού Κόμματος. Έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο. Δύο θέματα που ήδη αναφέρθηκαν. Σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Τζένι για τα πλεονεκτήματα περισσότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και των οργανώσεων Προστασία καταναλωτών στη χώρα μου, ασχολούμεθα πολύ με θέματα ανταγωνισμού και αυτό σημαίνει ότι υποτιμούμε συχνά θέματα προστασίας καταναλωτών. Νομίζω ότι το πολωνικό πρότυπο για περισσότερη συνεργασία χωρίς πλήρη ταύτιση των δύο θεμάτων θα μπορούσε να βοηθήσει. Βεβαίως, ε, ο ανταγωνισμός είναι προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη και αυτό που λέει ο κύριος Λούκε, ότι είναι κλειδί για διάφορα θέματα. Το δεύτερο. Το σημαντικό είναι να λειτουργεί καλύτερα η εσωτερική αγορά. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ αρμοδιοτήτων εθνικών αρχών ανταγωνισμού, αλλά αρκεί να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό για τις 28 εθνικές αρχές ανταγωνισμού. Ή μήπω θα έπρεπε να ε, θέσουμε το ερώτημα αυτό και στην 21η αρχή ανταγωνισμού, την Ευρωπαϊκή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θέλει κανείς άλλο τον λόγο πριν επιστρέψω στους ε, ομιλητές μας για να σχολιάσουν αυτά που είπατε. Α, παρακαλώ. Μία ερώτηση έχετε εσείς παρακαλώ. Πείτε μου και το όνομά σας. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πιερ από την εταιρεία booking.com. Κύριε Μόντι, Αναφερθήκατε στο θετικό παράδειγμα συνεργασία στην περίπτωση των επιγραμμικών ε, εταιρεών κρατήσεων ταξιδίων. Χαιρετίζουμε αυτή τη συνεργασία, αλλά υπάρχουν δύο προβλήματα. Ένα το αναφέρατε. Ένα κράτος μέλος έκανε κάτι εντελώς διαφορετικό, συγκεκριμένα η αρχή ανταγωνισμού του κράτου αυτού. Οπότε ποια είναι η κατάσταση. παραβιάζουμε τους στόχους της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Και επιπλέον, ο νομοθέτης λαμβάνει κάποιες αποφάσεις. Αλλά οι αποφάσεις δεν ρυθμίζουν το θέμα. Άρα η κατάσταση είναι λεπτή. Άρα το θέμα δεν είναι να, συνεργασ... να συντονίσουμε καλύτερα την εργασία των αρχών ανταγωνισμού, αλλά και μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού και των άλλων αρμόδιων αρχών για την ψηφιακή αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρο. Λίγουν λοιπόν οι ερωτήσεις και παρεμβάσεις ε, από την αίθουσα. Επαναρχόμεθα στους ομιλητές για καταληκτικές παρατηρήσεις. Τρία λεπτά παρακαλώ κάθε παρέμβαση. Και θα έλεγα να αντιστρέψουμε τη σειρά των αρχικών ε, παρουσιάσεων. Οπότε πρώτα θα πάρει το λόγο ο καθηγητής Μόντι. Τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με όλα, αλλά θα ασχοληθώ με ορισμένα. Πρώτα, η τελευταία ερώτηση για τις επιγραμμικές εταιρείες κρατήσεων. Ότι μια κρατική νομοθεσία ε, ακύρωσε τις αποφάσεις των αρχών ανταγωνισμού και σχετίζεται και με τι ρόλο παίζουν για τις κρατικές ε, επιδοτήσεις οι, αρχικές, οι αρχές ανταγωνισμού και τι ρόλο μπορούν να παίξουν για να δώσουν συμβουλές οι αρχές ανταγωνισμού για να υπάρξει σωστή νομοθέτηση, για να βελτιωθεί το οικονομικό όφελος. Κυρίως ασχολούμεθα με αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε ένα φετίχμα αυτό. Ο άλλος όμως ρόλος των αρχών ανταγωνισμού είναι να δίνουν συμβουλές ε, στις κυβερνήσεις ή να προτείνουν ε, νομοθετήματα. Στην Ιταλία για παράδειγμα, η Εθνική Αρχή επέκρινε την κυβέρνηση για ένα νομοθέτημα που μείωσε την ανταγωνιστικότητα της αγοράς ε, ε, ταξιδίων από το ίντερνετ. Ενώ καλύτερα θα ήταν να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός ή τουλάχιστον μέσω κάποια συζήτηση του δικτύου ανταγωνισμού για να βελτιωθεί ο ρόλος ε, ευαισθητοποίησης που έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Κάτι άλλο. Λέγεται ότι ο συγκεντρωτικός ε, ε, χαρακτήρας ε, είναι αρνητικός. Αλλά ξέρετε όλα τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν νομοθεσία που είναι ε, παράλληλη με την ενωσιακή νομοθεσία. Άρα δεν είναι θέμα εθελούσιου συγκεντρωτισμού. Είναι υποχρεωμένοι να ε, συντονίσουν την πολιτική τους. Και το τρίτο, οι ποινικέ ε, αποφάσεις ε, κάποιων εθνικών αρχών δείχνουν ότι δεν είναι η καλύτερη προσέγγιση αυτή. Γιατί οι ποινικέ αποφάσεις ε, καθιστούν την επίλυση μέσω, διαδικαστικών, με, μέσω διοικητικών διαδικασιών πιο δυσχερή. Ευχαριστώ κύριε Μόντι, καθηγητά Μόντι, λέει ο πρόεδρο, ο κύριος Κιζαράουσκας. Ευχαριστώ με την άδειά σα Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο μου στα δεξιά, τον κύριο Ζενή, ο οποίο ε, βιάζεται γιατί πρέπει να πάρει το τρένο να γυρίσει. Βεβαίω, καθηγητά Ζενή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χρησιμοποιήστε το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Ετέθηξαν πολλά ερωτήματα και δεν μπορώ να τα απαντήσω όλα, ιδιαίτερα εκείνα που αφορούσαν την Ιρλανδική Αρχή Ανταγωνισμού, εγώ θα αναφέρω το εξή. Είναι δύσκολο να έχουμε ένα κοινό πρότυπο. Και αυτό γιατί διαφέρει, διαφέρουν οι μορφές που παίρνουν και το μοντέλο που ακολουθείται ε, όσον αφορά τις αρχές ανταγωνισμού σε κάθε χώρα. Δηλαδή, εάν πρόκειται για διαδικασία διοικητική ή ποινική. Αυτό ε, αλλάζει κατά πολύ τα πράγματα. Γι' αυτό είπα ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το ίδιο μοντέλο παντού στην Ευρώπη και κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να αποφασίζει εκείνο ποιο μοντέλο θέλει να ακολουθήσει. Η επιβολή ε, ποινικών κυρώσεων, δηλαδή το να ακολουθείτε μια ποινική διαδικασία, βεβαίω αυξάνει ε, το κόστο, ε, κάνει τη διερεύνηση των υποθέσεων πιο δυσχερή, γιατί εκεί το βάρο τη απόδειξη είναι πιο αυστηρό και πιο περίπλοκο συνήθω το σύστημα από τις ε, διοικητικέ κυρώσει. Τώρα όσον αφορά τους ε, υπαλλήλου τη Επιτροπή, οι οποίοι πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα και ξαναγυρνούν και εργάζονται στι ίδιε υποθέσει. Εδώ το ζήτημα είναι ευαίσθητο. Δεν έχει ε, δεν έχουν συζητηθεί διεξοδικά κανόνες, για παράδειγμα κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει μια περίοδος ε, κατά την οποία δεν θα επιτρέπεται ε, κάποιος να εργάζεται σε τέτοιου τύπου αρχές, επιστρέφοντας από μια άλλη σχετική θέση. Είναι το μοντέλο που έχει ακολουθήσει η Γερμανία, για παράδειγμα. Εδώ όμως, όπως είχα πει, υπάρχουν δύο ζητήματα ανεξαρτησίας. Πρώτον, το θεσμικό πλαίσιο, η ανεξαρτησία της αρχής ανταγωνισμού που επιβάλλεται στον νόμο και αφετέρου το κατά πόσον η ίδια η αρχή ανταγωνισμού έχει τη βούληση να διαφυλάται την ανεξαρτησία της, να εργάζεται ανεξάρτητα. Πιστεύω ότι είναι πιο δόκιμο να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ μιας ε, ξεχωριστή αρχή ανταγωνισμού και μια ξεχωριστή αρχή για τα δικαιώματα του καταναλωτή, αντί να συγχωνεύονται αυτέ οι δύο αρχέ. Όπω σα είπα, υπάρχουν ε, πλεονεκτήματα και αμενιοκτήματα, όποια και από τι δύο λύσει και αν επιλέξει κανεί, δηλαδή αν τη συγχωνεύσει ή όχι. Ε, γι' αυτό δεν μπορώ να πω ότι ένα μία από τι δύο επιλογέ είναι η καλύτερη, εξαρτάται από την κατάσταση σε κάθε κράτο. Πράγματι σε κάποιες χώρες ίσως να είναι καλύτερα να υπάρχουν δύο ξεχωριστές αρχές που να συνεργάζονται. Υπάρχει επίσης και μια άλλη πιθανότητα, την έχουμε δει σε χώρες εκτός Ευρώπης, ε, να υπάρχουν δύο αρχές οι οποίες να αποτελούν τμήματα του ιδίου οργανισμού ή του ιδίου θεσμικού οργάνου και παρόλα αυτά να μην συνεργάζονται. όσον αφορά τις, τα θεσμικά ζητήματα των διώξεων. Αναφερθήκαμε μόνο σε εκείνα τα, τα, τις πτυχές του θεσμικής ε, λειτουργίας που ε, έχουν επιπτώσει στην αποτελεσματικότητα. Πρώτον, μπορεί κανείς να φροντίσει να υπάρχει ε, διαχωρισμός μεταξύ των ε, δικαστών και των εισαγγελέων έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η ορθή επεξέταση της, ε, της υπόθεσης. όποιο μοντέλο και αν επιλέξει κανείς δηλαδή για το εάν η αρχή θα είναι συγχωνεμένη, αν θα υπάρχουν δύο αρχές, έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Έχουν υπάρξει και καινοτόμες προτάσεις για το πώς μπορούν να συνδυαστούν διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης το πρόβλημα με μια αυτόνομη πηγή χρηματοδότηση συχνά είναι ότι δεν ε, συναπάται με το φόρτο εργασία τη αρχή, Το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα αν κάποια στιγμή ξαφνικά η αρχή πρέπει να ασχοληθεί ε, με πολλές υποθέσεις, αν υπάρχουν για παράδειγμα πολλέ συγχωνεύσεις εταιριών. Γι' αυτό χρειάζονται και, άλλε και άλλες πηγές χρηματοδότησης, ε, όπως για παράδειγμα το μοντέλο της Ιταλίας ή το μοντέλο της Πορτογαλίας, που έχουν και σταθερές αυτόνομες πηγές χρηματοδότησης και ε, άλλες πηγές που σχετίζονται με τα πρόστιμα που επιβάλλει η αρχή έτσι ώστε τελικά ε, να έχει την χρηματοδοτική αυτονομία η αρχή που χρειάζεται. Ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Κεσεράουσκος για τρία λεπτά. Ευχαριστώ όσον αφορά την θεσμική ανεξαρτησία και την προσωπική ανεξαρτησία. Το πρώτο είπαμε ότι μπορεί να ε, τον γεθεί το δίκαιο νόμος, το δεύτερο ε, δυσκολότερο. Αλλά μπορεί αυτή η αρχή ανταγωνισμού να του καθιστά τους πάντες ότι υπάρχουν εγγύησεις ότι η υπάλληλοι είναι ανεξαρτητή, Αλλά δεν μπορεί να γίνει το αντίστροφο δηλαδή τα πρόσωπα να πείσουν για την υπηρεσία. Οπότε θα πρέπει να δούμε κατά πόσον είναι δυνατόν να, να αναμειχθεί ή όχι το κράτος. Επίσης είπαμε τι γίνεται με σύγκρουση συμφερόντων, τι, τι, τι κάνουν οι αξιωματούχοι όταν ε, λήξει η θητεία τους. Το θέμα αυτό εκρεμεί. Δεν έχει λυθεί σε πολλές χώρες. Στην Λιθουανία έχουμε ένα έτος ε, κατά το οποίο παγώνει στα διαδρομία του αξιωματούχου. Και βέβαια αυτό είναι αντικίνητρο. Γιατί δίνεται αποζημίωση με τη μόνο ενό μηνό. Άρα κανεί δεν θέλει να πάει να γίνει αξιωματούχο. Και από την άλλη μεριά, επειδή είναι τόσο εξειδικευμένο το αντικείμενο, όταν λήξει η θητεία δεν μπορεί να βρει κανεί άλλη δουλειά. Τώρα όσον αφορά την χρηματοδότηση πάλι παραπέμπουμε ε, στο κύριο Ζενή. Τα λεγόμενα υπάρχουν πολλά παραδείγματα στη χώρα μας όπου είχαμε κάποια νομοσχέδια που προσπαθήσαμε να περάσουμε και η χρηματοδότηση θα γινόταν από κάποιες χρηματικές ποινές, όπως ακριβώς είναι και στην Ιταλία. Τέλος, λέμε για ένα αποτελεσματικό σύστημα σε σχέση με την αποτελεσματική αρχή. Τι θέλουμε. Και τα δύο τα θέλουμε. Γιατί η αποτελεσματική υπηρεσία δεν μπορεί να ε, φτιάξει αναγκαστικά αναγκαστικό σύστημα αλλά και το σύστημα δεν μπορεί να συγκροτήσει μια ε, αποτελεσματική υπηρεσία από μόνο του. Άρα και τα δύο τα θέλουμε. Κύριε Γκόγεν, σας ευχαριστώ για να σα πω δύο λόγια όσον αφορά την συνεργασία με το κράτος όπως ε, ρωτήθηκε. Δεν υπάρχει κανόνα για το να πρέπει η ίδια αρχή να ρυθμίζει τον ανταγωνισμό και τα σύμφωνα των καταναλωτών. Σαν να κάθε χώρα. Αλλά βέβαια θα υπάρχουν διαφορετικέ υπηρεσίε, θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ του. Γιατί υπάρχουν πολλέ επικαλύψει, πολλά κοινά μέτωπα. Ε, χρειάζεται μια υπηρεσία την εμπειρία τη άλλη. Αλλά θέλω να σα πω, μην κολλάτε μόνο στο θέμα τη συνεργασία αυτών των δύο αρχών. Γιατί υπάρχουν και άλλε αρχέ που μπορούν να βοηθήσουν την αποτελεσματικότητα των αρχών του ανταγωνισμού. Γιατί είναι τόσε πολλέ πληροφορίε που μπορούν να, να ε, διαβαστούν. Ας πούμε έχουμε την υπηρεσία προστασίας των δεδομένων, ε, έχουμε τις ρυθμιστικές αρχές για επικοινωνία, για φάρμακα κλπ. Άρα χρειάζεται διάλογος, επαφή όλων αυτών των υπηρεσιών. Και έτσι να ξεδαστούν οι προτεραιότητες να είναι οι και αυτό εξοικονομεί και πόρους. Ε, γιατί κανείς δεν χρειάζεται να προσπαθείς για να επισημάνει αυτό που διαφορά. Τώρα, όσον αφορά ομαδικές ε, αγωγές, ναι, αυτό είναι ένα μέσον αποτελεσματικό. Και θα πρέπει κάτι τέτοιο να αναπτυχθεί. Δεν είμαι ειδική για αυτές τις ε, αγωγές, αλλά νομίζω όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου στον ιδιωτικό τομέα ότι υπάρχει κάποια οδηγία Επομένως, μπορούν οι φορείς των καταναλωτών να προσφέρουν ομαδικές ε, αγωγές. Ευχαριστώ πολύ. Και για να λήξουμε το γύρο καταληκτικών παρατηρήσεων των ομιλητών, η κυρία Φερνάντες, τρία λεπτά. Ευχαριστικό, τα περισσότερα έχουν ήδη υποθεί. Να μιλήσω για την ενδεχόμενη εκ νέου συγκεντρωτική τάση αυτής της προσπάθειας και αν είναι κατάλληλη στιγμή. Όταν ε, έλεγα ότι είμαι υπέρ ε, νέας εναρμονισμένης νομοθεσίας, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι χρειαζόμαστε ένα ενιαίο σύνολο δικαιωμάτων για τις εταιρείες παντού στην Ευρώπη. Γιατί τώρα σε πολλά κράτη-μέλη δεν υπάρχουν ε, προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις για θέματα των άρθρων 101-102 στην Ισπανία. Υπάρχουν σαφείς προθεσμίες, 18 μήνες για παράδειγμα είναι εκεί. Οι επιχειρήσεις θα ήθελαν να υπάρχει ενιαία προθεσμία για να ξέρουν μέχρι πότε θα μπορούν να έχουν την απόφαση για μια διαδικασία για τελειώσει. Υπάρχει κόστος, υπάρχει αβεβαιότητα, είναι κακό για τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι τομεί, για παράδειγμα διαδικασίες δικονομικά, σε πολλού άλλους τομεί. οι δυνατότητε που έχουν οι αρχές ε, να υποβαθμίσουν κάποιες επιχειρήσεις. Όλα αυτά ποικίλουν από χώρα σε χώρα, άρα οι επιχειρήσεις ε, έχουν πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν ε, ελάχιστα δικαιώματα στα οποία να μπορούν να βασιστούν οι εταιρείε για να μπορούν να λειτουργήσουν ε, παντού στην Ευρώπη και για να κρυθούν με παρόμοιο τρόπο. Ταυτόσιμο θα έλεγα. Συμφωνώ με τον καθηγητή κύριο Μόντι και το είπα ήδη δεν ε, παίζουν επαρκώς το ρόλο ε, να προωθήσουν ε, την ευαισθητοποίηση για θέματα ανταγωνισμού οι εθνικές αρχές. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να το κάνουν περισσότερο. Δεν είναι μόνο η δυνατότητα να δώσουν νομοδοτήσεις, να προτείνουν νομοθετήματα, να κάνουν εκθέσεις για να βοηθήσει τον ανταγωνισμό, το νομοθετικό πλαίσιο παντού στην Ευρώπη. Οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού θα πρέπει να έχουν δυνατότητα να προσφύγουν και στο δικαστήριο για να αμφισβητήσουν νομοθετήματα που θίγουν τους κανόνες ανταγωνισμού. Αυτή είναι η εγγύηση ομογενοποίησης του πλαισίου στην Ευρώπη. Οι αρχές αυτές θα έπρεπε να προωθούν ε, τον ανταγωνισμό και σε νομοθετικό επίπεδο. Και κάτι ακόμη η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών, ιδιαίτερα στα πλαίσια του δικτύου, που είναι σημαντική δυνατότητα για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Πρέπει να υπάρχει και διαφάνεια σε αυτή τη συνεργασία. Γιατί θα παίξει και αποτρεπτικό ρόλο. Αν οι εταιρείε ξέρουν ότι συνεργάζονται αυτές οι αρχές, τότε οπωσδήποτε θα αποφύγουν τις παραβιάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Οπότε κλείνουμε το πρώτο γύρο παρουσιάσεων, το πρώτο πάνελ. Νομίζω ότι οι παρουσιάσεις αλλά και οι παρεμβάσεις ε, από τους παρευρισκόμενους ε, έδειξαν πολλά θέματα που αναφέρθηκαν και στη δημόσια διαβούλευση. Το θέμα της ανεξαρτησίας των εθνικών αρχών ανταγωνισμού τονίστηκε ότι είναι ζωτική σημασία. και το ανέφεραν πολλοί από διάφορες πλευρές. Επίσης ε, η σημασία επάρκεια σπόρων. Πολλά υπόθηκαν και για την ε, ανεξαρτησία και αυτονομία του προπολογισμού και αναφέρθηκαν και οι διαφορές μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού και της χρηματοδότησής τους, γιατί πολλές φορές αυτές οι προσπάθειες επιβολής του δικαίου ανταγωνισμού μπορεί να αφορούν κρατικούς φορείς, το κράτος, το οποίο δίνει για τον προπολογισμό. Ε, παρέχει τον προπολογισμό. Η συνεργασία μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού αναφέρθηκαν και το θέμα της σωστής ισορροπίας μεταξύ ε, διαδικαστικών εγγυήσεων και σωστής εφαρμογής του νόμου. Όλα αυτά τα, θέματα αναφέρθηκαν και στη δημόσια διαβούλευση. Η Κομισιόν σημειώνει προσεκτικά όλα όσα υπόθηκαν. Επίσης, αναφέρθηκαν και άλλα θέματα που είναι ευρύτερα και αυτά τα σημειώνουμε προσεκτικά. Να αναφέρω ορισμένα μόνο. Ο συντονισμός ε, στα πλαίσια του δικτύου σχετίζεται με τα θέματα της δημόσιας διαβούλευσης γιατί όσο πιο εξοπλισμένες και αποτελεσματικές είναι οι αρχές ανταγωνισμού τόσο καλύτερα μπορούν να συντονιστούν. Αλλά θέλω να τονίσω ότι το θέμα του συντονισμού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού είναι ένα θέμα που το συζητά συνεχώς η Επιτροπή με τις Εθνικές Αρχές και εργαζόμεθα για τη βελτίωσή του. Το θέμα των ε, κρατικών επιδοτήσεων και βοηθειών εφήγει. Βέβαια είναι διαφορετική κατάσταση ε, από την κατάσταση καταπολέμησης των καρτέλ, γιατί εδώ οι στρεβλώσεις προκύπτουν από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Και αποκλειστική αρμοδιότητα για την εφαρμογή των κανόνων των, για την κρατική βοήθεια είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά αυτό δεν αποκλείει περισσότερες δυνατότητες ε, δράσης στον τομέα αυτό για τις εθνικές αρχές, ιδιαίτερα στα πλαίσια του εξυγχρονισμού των κανόνων για την κρατική βοήθεια που προσπαθεί να εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια η Κομισιόν, αλλά είναι δύο διαφορετικά συστήματα. Άρα δεν μπορούν να ενοποιηθούν πλήρως. Και τώρα για την επιβολή του νόμου σε περιπτώσεις ε, φυσικών προσώπων. Η σχετική οδηγία, υπενθυμίζω, πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι τον ε, προσεχή Δεκέμβριο. Τότε λίγη προθεσμία. Νομίζω λοιπόν ότι το πάνελ κάλυψε αναλυτικά τα θέματα καταμερισμού εργασίας μεταξύ του ευρωπαϊκού και του εθνικού επίπεδου για τα θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας αντιτράστ με πιο αποτελεσματικό και ισότιμο τρόπο. Και αυτό έχει να κάνει και με το πόσο πολιτικά ευαίσθητο είναι το θέμα αυτό. Τι συζητάμε σήμερα. Δεν θέλουμε να περάσουν αρμοδιότητες από το εθνικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αντίθετα να γίνει σωστός καταμορισμός εργασίας μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού επίπεδου με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ιδίω σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ λοιπόν τους πέντε ομιλητές μας, θερμότατα, για την παρουσία τους, για την προπαρασκευή τους, για τις παρεμβάσεις τους και ευχαριστώ και όλους όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση και ε, να δώσω και πάλι την Προεδρία στον Πρόεδρο Γκουαλτιέρη. Σας ευχαριστώ. Νομίζω το πρώτο πανέλ ομιλητών ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον και τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο που και εκείνο θα ασχοληθεί με ένα κρίσιμη σημασία θέματα, θέμα το ζήτημα του πώς θα γίνει αυτός ο καταρρομεριασμός εργασίας πιο αποτελεσματικός είναι το θέμα των προγραμμάτων επίοικειας και οι κυρώσεις στα κράτη-μέλη όταν εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τον ανταγωνισμό. Τα προγράμματα επί προβλέπονται στους ευρωπαϊκούς κανόνες ε, για τον ανταγωνισμό. Αλλά όταν διαπιστώνουμε ότι τα πρόστιμα ε, εφαρμόζονται σε, στα, επιβάλλονται μάλλον στα κράτη-μέλη, υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε κάποια ε, κράτη-μέλη πρόστιμα μπορούν να επιβάλλουν μόνο τα δικαστήρια, ενώ σε άλλα κράτη-μέλη ε, μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα και οι ίδιε οι αρχές ανταγωνισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει ένα ανώτατο όριο στο ποσό του προστίμου και σε πολλές περιπτώσεις επίσης τα πρόστιμα υπολογίζονται διαφορετικά. Όλα αυτά έχουν ως, αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί ένα σύστημα με βάση το οποίο θα υπάρχει ένα μέγιστο όριο του 10% ε, του κύκλου εργασιών. Επίσης, οι ποινικέ διώξεις δεν είναι κάτι το οποίο ε, συμβαίνει συχνά. Τα προγράμματα επί σε γενικές γραμμές εναρμονίζονται με τις ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως το θέμα είναι ε, εάν αυτά τα προγράμματα επί τελικά ε, εφαρμόζονται διαφορετικά από κάθε κράτος μέλος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να διερευνήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Προσπαθήσαμε να έχουμε εκπροσώπους από πολλές διαφορετικές πτυχές, εκπροσώπους των επιχειρήσεων, των ε, γραφείων συμβούλων, ε, του δικαστικού σώματος, των ε, επιτροπών καταναλωτών κτλ. Θα δώσω το λόγο στον πρώτο μας ομιλητή, ο κύριος Παύλο Μπάρος, μέλος της ομάδας των εργοδοτών στην ΕΟΚΕ στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Ε, ως εκπρόσωπος των ενώσεων επιχειρήσεων. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ, θα μιλήσω πορτογαλικά. Εκ μέρου τη Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνική Επιτροπής θα ήθελα να ευχα... σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση οι ομιλητές από ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισαν την ε, σημασία της κοινωνίας των πολιτών και η ΟΚΕ εκπροσωπεί ακριβώς αυτή την κοινωνία των πολιτών. Τα τελευταία χρόνια έχουμε διαπιστώσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει όλο και πιο φιλόδοξες πρωτοβουλίες στον τομέα της αντιμονοπολιακής νομοθεσίας, πιο συγκεκριμένα μέτρα, και πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αφορούν τομείς ε, της οικονομίας. στοχεύοντας η καλύτερη ε, προστασία του καταναλωτή και βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Η έκθεση ε, προτείνει τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να ξεκινήσει να δραστηριοποιείται περισσότερο. Όμως, η δικιά μας εμπειρία την πλευρά των εργοδοτών που εκπροσωπούνται στην ΕΟΚΕ και εμείς εκπροσωπούμε αυτούς που πραγματικά ε, επιχειρούν ε, στις διάφορες χώρες. Μας έχει επιτρέψει λοιπόν αυτό να έχουμε μια πιο ε, ρεαλιστική προσέγγιση και να έχουμε τη δυνατότητα να συγκεράζουμε αντικρουόμενα συμφέροντα και αντικρουόμενες απόψεις. Θα σας δώσω λοιπόν κάποια στοιχεία και κάποιες πληροφορίες που ε, έχουμε συλλέξει ως παράδειγμα από την Πορτογαλία. Το 2013 υπήρχε μια γενική διεύθυνση ε, σε ένα Υπουργείο, αρμόδια για ζητήματα ανταγωνισμού. Ε, δημιουργήθηκε το 2013 ένα εντελώ καινούριο νομικό πλαίσιο, το οποίο διασφάλιζε καλύτερα την ανεξαρτησία. Και στα τρία χρόνια που μεσολάβησαν είδαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις. Δημιουργήθηκαν ρυθμιστικές αρχές, δημιουργήθηκε ένα εξειδικευμένο δικαστήριο ε, για ζητήματα ανταγωνισμού. Βελτιώθηκε λοιπόν συνολικά το θεσμικό πλαίσιο της Πορτογαλίας με βάση τις βέλτιστες πρακτικές που είδαμε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι καταφέραμε να δημιουργήσουμε και ένα σύστημα προγραμμάτων ευηγικίας που στην Πορτογαλία μας επέτρεψε να καταπολεμήσουμε καρτέλ. 19 υποθέσεις ξεκίνησαν να διαρευνώνται από το 2013. Οι ε, νέα αφορούσαν καρτέλ, οι 5 κατάχρηση δεσπόζουσα θέσεις και μάλιστα μία από αυτές οδήγησε σε μία ε, επιβολή σημαντικής ποινής, σημαντικής κύρωσης στην εταιρεία, τη δημόσια εταιρεία φυσικού αερίου. Το σχετικό πρόστιμο περίπου 20 εκατομμύρια ε, ευρώ. Υπήρξε επίση και μια σημαντική πηγή χρηματοδότηση για την Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού. Ένα άλλο ζήτημα που εξετάστηκε ήταν τα καρτέλ που δραστηριοποιούνταν στον ε, χώρο ε, των, της, της, των για τα σχολεία. μια άλλη υπόθεση η οποία διερευνήθηκε ήταν τα ενυπόθηκα δάνεια και οι πρακτικές που ακολουθούσαν οι διάφορες τράπεζες σε αυτά. Και στις δύο αυτές τελευταίες δύο υποθέσεις που ανέφερα χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα επί για την απόκτηση περισσότερων στοιχείων. Καθώς με την πάροδο του χρόνου τα προγράμματα επίκαιας έχουν γίνει πιο προβλέψιμα. Ε, γίνεται πιο ξεκάθαρο πώς μπορεί μια επιχείρηση να αξιοποιήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα επίκαιας αποφεύγοντας ε, τις ε, κυρώσεις και διευκολύνοντας την έρευνα με νομοθεσία του 2012 ε, διευκρινίστηκε καλύτερα τι συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και πώς ε, υπολογίζεται, πώς ερευνάται εάν υπάρχει οικονομική σχέση εξάρτησης μεταξύ δύο εταιριών. Θέλω να σταθώ λίγο περισσότερο στο πώς λειτουργεί το σύστημα ε, των προγραμμάτων στην, στην Πορτογαλία. έχουν επωφεληθεί από αυτό μέλη διοικητικών συμβουλίων, ελεγκτικές εταιρείες. Όταν μια ε, επιχείρηση η οποία ερευνά το για ε, παραβίαση της νομοθεσίας για το ανταγωνισμό ε, συνεργαστεί πλήρως με την αρχή ανταγωνισμού και μας δώσει στοιχεία για καρτέλ, τότε δεν της επιβάλλεται καμία κύρωση. αλλά προβλέπεται ρητό στο νόμο ότι αυτό σημαίνει ότι θα μας ε, παρέχει όλα τα στοιχεία που τις ε, ζητούνται, ε, θα υπάρχει πλήρη συνεργασία. Συνοψίζοντας, έχουμε δει ότι το πρόγραμμα επίγειας ήταν αποτελεσματικό. Εμείς έχουμε ένα όριο ε, στο, στο, στο, στο στην ανώτατη κύρωση που μπορεί να επιβληθεί στο 10% του κύκλου εργασιών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Η κυρία Έντοτσον που είναι δικαστής στο διοικητικό εφετείο. Και το 2015 ε, ασχολείται με το θέμα μας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, να σας πω για την σουηδική εμπειρία. Θεωρούμε τα προοδευτική χώρα. Όμως, όσο αφορά το σήμερα συζητούμενο θέμα, είμαστε ουραγοί. Στην Σουηδία θα πρέπει πρώτα να κριθεί κατά πόσον η αρχή επί του ανταγωνισμού θα μπορεί να αποφασίζει για τις χρηματικές ποινές και πρόστιμα. Και έχουμε την έκθεση του 2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την νομοθεσία αντιτράστη. Ο καθένας έχει ένα μοντέλο. Και εμείς, σε κάποια κρατημέλη μάλλον, η αρχή του ανταγωνισμού έρευνα τις περιπτώσεις παραβίαση του δικαίου ανταγωνισμού Φιλανδία, Ιρλανδία και Αυστρία έχουν συστήματα που μοιάζουν με το δικό μας. Οπότε κάποια μέλουσα ε, η κοινωνική νομοθεσία θα πρέπει να αποφασίσει για το κατά πόσο αρχή του ανταγωνισμού θα έχει τέτοιες εξουσίες έρευνας. Οπότε και εμείς θα πρέπει να δούμε αν θα αλλάξει το σύστημά μας, το οποίο ισχύει από το 1953. Ευτυχώς η κυβέρνηση ε, από μόνη της έχει αρχίσει να τα σκέφτεται κατά αυτόν τον τρόπο. Πέρσι είχαμε κάποια κυβερνητική επιτροπή η οποία αναβάθμισε την αρχή ανταγωνισμού όσον αφορά τις αποφάσεις που μπορεί να πάρει. Και θα υπάρξει και κάποια έκθεση που θα δημοσιοποιηθεί τον Ιούνιο. Για να δούμε τώρα κάποια θέματα που μας απασχολούν στη Σουηδία, αλλά έχουν και σχέση με τη σημερινή μας ακρόαση. Κράτος δικαίου, αποτελεσματικότητα και εναρμόνιση. Πρώτα-πρώτα, οι επιχειρήσεις αλλά και οι πολιτικοί συζητούν αν θα πρέπει α, να πάμε από το διοικητικό ε, σε ένα άλλο ε, πρότυπο. Και θα πρέπει όμως να δούμε κατά πόσον το πρώτο που θα ακολουθούμε συνάδει προς τον χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί ζητούμε να μας μιμηθούν κάποια κράτη-μέλη. Αλλά αυτό δεν συνέβη, άρα θα πρέπει να αναθεωρήσουμε. Πάντως Υπάρχουν κάποια επιχειρήματα αλλαγή του πρότυπου τα οποία έχουν πιάσει τόπο και υπάρχει κάποια έκθεση που έχω συντάξει σχετικά. Επομένως, συντάξαμε, δεν έχω μόνο στα, στα μία μελέτη όπου έχουμε τη γνώμη 26 προσώπων από τον ε, νομικό κόσμο. Και αυτό που προκύπτει είναι στο ότι υπάρχει δυσπιστία μεταξύ νομικών και της αρχής ανταγωνισμού. Η αρχή ανταγωνισμού θεωρεί ότι παρελκύουν τις έρευνες οι δικηγόροι. Αλλά και οι δικηγόροι δεν εμπιστεύονται όσον αφορά τη λήψη κάποιες απόφασεις στην αρχή ανταγωνισμού. Άλλη βέβαια είναι η σχέση των νομικών προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε η αλλαγή του προτύπου θα, θα μας οδηγούσε στο να πάει κανείς στη φυλακή απευθείας από τον εισαγγελέα. Για την αποτελεσματικότητα τώρα. Στην έκθεσή μου προσπαθώ να αναλύσω το γιατί είναι πιο αποτελεσματικό το διοικητικό πρότυπο. Παρά το δικαστικό. Έχουμε 28 αρχές συνταγωνισμού και θα πρέπει να το κάνει αυτό το ίδιο μοντέλο, το εφαρμόζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως αυτά που σήμερα συζητήσαμε θα τα λάβουμε υπόψη μας για το τι θα κάνουμε στην Σουηδία. Δεν ξέρω τελικά τι θα κρυθεί και τι θα αποφασίσει το Κοινοβούλιο και η κυβέρνησή μας. Γιατί πάντοτε ισχύει το ότι όταν κάτι λειτουργεί θα πρέπει να το πειράζει κανείς. Πάντω σημασία έχει το κακό υπάρχει εμπιστοσύνη προ ένα ισχύον σύστημα. Είπαμε εναρμόνιση των ερευνητικών αρμοδιοτήτων και να έχουν όλε οι εθνικέ αρχέ τι ίδιε αρμοδιότητε, αυτέ που είχε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό εννοούμε. Ή θέλουμε ομοιογένεια με άλλες αρμοδιότητες. Έχει δίκιο εδώ η θελουμε ομοιογενεια με αλλε αρμοδιοτητε εχει δικιο εδω η επιτροπη που λέγεται την εξισορρόπηση των ε, συμφερόντων, δηλαδή από τη μια μεριά το κράτος δικαίου και από την άλλη μεριά τις οικονομικές εγγύησεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γκουίντο Λουμπράνο, ο οποίος είναι αναπληρωτής διευθυντής της Business Europe. Είναι συντονιστής για την ε, νομική πλευρά της ενιαίας αγοράς και είναι αρμόδιος απευθείας για την πολιτική ανταγωνισμού και τις ε, κρατικές βοήθειες και για ψηφιακά οικονομικά θέματα αντιπρόεδρος επίσης της ομάδας εργασίας για θέματα ανταγωνισμού του οργανισμού Business Europe. Έχει εργαστεί ως εξωτερικός εμπειρογνώμων για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Κύριος Μπράνο, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταρχάς θέλω να τονίσω ότι η οργάνωσή μας είναι Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων. Άρα συμμετέχουμε γιατί μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η συζήτηση και ενδεχόμενα είμαστε και εναγόμενοι σε ορισμένε τέτοιες υποθέσεις. Και έχουμε και ένα ρόλο που σχετίζεται με τον ανταγωνισμό, ως εναγόμενοι λοιπόν, ενδεχόμενα και ως αγωγή, φυσική, πολιτική αγωγή και θύματα. Άρα θέλουμε να υπάρχει ένα πολύ ρωμαλαίο και δίκαιο σύστημα επιβολής της πολιτικής ανταγωνισμού. Ο εξυγχρονισμός του 2003 σκόπευε να εφαρμόζεται το δίκαιο ανταγωνισμού από τις εθνικές αρχές γιατί θεωρείται ότι ήταν ε, ο καλύτερος φορέας για να το κάνει αλλά παράλληλα η Κομισιόν θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να ασχολείται με θέματα που έχουν περισσότερες επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός ο εξυγχρονισμός δεν ήθελε να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στην εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού για τις κυρώσεις, ε, τα ένδικα μέσα, τις δυνατότητες ε, προσφυγής κτλ. Έφεσης καλύτερα. Ανάλογα με το εάν ε, η αρχή που θα εφήρμοζε το δίκαιο ανταγωνισμού είναι εθνική ή κομισιόν. Βλέπουμε τη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε η κομισιόν. Βεβαίω είναι πολύ σημαντική η στόχη αυτή και συμμεριζόμεθα τους στόχους αυτούς. Θέλουμε να υπάρξει περισσότερη ενοποίηση στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς, ακριβώς και για τον ανταγωνισμό. Για τον ανταγωνισμό. Και επίσης και ανεξαρτησία είναι θέμα πολύ λεπτό, σημαντικό για τις επιχειρήσεις. Αλλά είναι κάπως ε, πιο ιδεαλιστική η προσέγγιση, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει μεγάλος κατακαιρματισμός ο επιχειρηματικό κόσμος θεωρεί ότι οι περισσότερες αρχές ανταγωνισμού τα πάνε πολύ καλά. Έχουν πολύ υψηλό επίπεδο σωστή ε, σωστή Για παράδειγμα, οι δηλώσει ε, αντιρρήσεων είναι κάτι το οποίο οι δικηγόροι το θεωρούν δύσκολο. Και ορισμένα μέλη μας πρόσφατα μας είπαν ότι σε κάποιες χώρες της Κεντρική Ευρώπη λίγο πριν ε, το Πάσχα, μία εθνική αρχή ζητάει από μια μικρή επιχείρηση όλα τα έγγραφα που διαθέτει, όλα, κυριολεκτικά, σε μια εβδομάδα. Ε, έγινε κάτι τέτοιο δηλαδή. Κάτι που ήταν αδύνατον, χωρίς καμία δυνατότητα παράταση. Μόνο και μόνο η συλλογή όλων των εγγράφων από όλου του εργαζόμενου σε αυτή την εταιρεία χρειάζεται εβδομάδε. Γι' αυτό λοιπόν δώσαμε αυτές τις απαντήσεις και λίγο πιο επιφυλακτικές ε, σε αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης. Η πρώτη μας απάντηση είναι ότι όλες οι αρχές, όλες οι εθνικές αρχές πρέπει να σέβονται περισσότερο την ορθή διαδικασία σε όλες τις χώρες για το ποιοι συμμετέχουν. Αν θα πρέπει να είναι οι εναγόμενοι, οι ενάγοντες, οι καταναλωτές, το θέμα είναι εάν θα είναι κάποια εθνική αρχή ή η οι κομισιον Χρειάζονται οι εθνικές αρχές περισσότερες αρμοδιότητες για να καθορίζουν αυστηρότερες ποινές. Εμείς θεωρούμε όχι. Στις περισσότερες δικαιοδοσίες είναι παρόμοιες οι κυρώσεις. Με βάση αυτό το 10% του κύκλου εργασιών ως ανώτατο όριο. Και τα δικονομικά δικαιώματα, βεβαίως, είναι ανησυχία για τον επιχειρηματικό κόσμο. Να μην υπάρχουν διακρίσεις, να υπάρχει δυνατότητα να ακουστούν, να ε, λήγουν διαδικασίες σύντομα, να είναι ανάλο, ανάλογες, να, να τηρείται η αναλογικότητα. Και θεωρούμε ότι το σουδικό σύστημα είναι ιδιαίτερα πεφωτισμένο. Έχει βέβαια κάποιες αδυναμίες αλλά από την πλευρά της στήρησης της νομιμότητας και των διαδικασιών είναι πολύ καλό παράδειγμα. Και τα συμπεράσματά μας είναι ότι θα θέλαμε η διαδικασία αυτή να καταλήξει σε μια δέσμευση όλων των εθνικών αρχών να σέβονται αυστηρά τις βέλτιστες πρακτικές που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως τις καθόρισε το 2011 για τις δικές της διαδικασίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μην είναι τέλειες αλλά είναι πολύ καλό παράδειγμα αυτού που θα ήθελε ο επιχειρηματικός κόσμος να είναι το επίπεδο των ε, διαδικαστικών εγγύσεων. Κάτι άλλο. Τα προγράμματα επίοικειας. Ναι, ναι, είναι ζωτικό στην περίπτωση των καρτέλ. Ε, συμφωνεί ο επιχειρηματικός κόσμος, αλλά σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα. Ένα σαφές μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε είναι να υπάρχει ένα σύστημα με δείκτες. Marker system. Ότι αν ε, κάνεις αίτηση επί και είσαι ο πρώτος ο οποίος παραδέχεται την ε, παράβαση, τότε να μην κινδυνεύεις ε, από τα διαφορετικά εθνικά συστήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Θα περάσουμε στην επόμενη ομιλήτρια, η Σόλτιν Κόκκιν, συγγνώμη, ε, πρόεδρος της Ιρλανδικής Αρχής για τον Ανταγωνισμό και την Προστασία του Καταναλωτή. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Η Ιρλανδία είναι μια μικρή χώρα και έχει ανοιχτή οικονομία, το οποίο σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός είναι πολύ σημαντικός για εκείνη, για την επιτυχία της οικονομίας της, για τις εξαγωγές της, ίσως περισσότερο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Προσπαθούμε λοιπόν η οικονομία να παραμένει ανοιχτή, να δίνουμε τη δυνατότητα σε νέες ε, επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται και τις παλαιότερες ευρεωμένες να συνεχίζουν να το πράττουν η στρέβλωση του ανταγωνισμού μπορεί να δημιουργηθεί είτε όταν υπάρχει μία εταιρεία που έχει δεσπόδουσα θέση, είτε όταν μία ομάδα επιχειρήσεων δημιουργήσει καρτέλ. Ο ανταγωνισμός λοιπόν είναι κάτι το οποίο αφορά και τις μικρές και τις μεγάλες επιχειρήσεις, το οποίο σημαίνει ότι οι επιβληθήσεις ποινές, οι επιβαλλόμενες ποινές θα πρέπει να προσαρμόζονται στο μέγεθος της εταιρεία. Η δημιουργία από την άλλη ενός καρτέλ έχει δυσμενείς επιπτώσεις στους, ιδίως στους καταναλωτές. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, για αυτόν τον λόγο, πιστεύω ότι χρειάζονται και ποινικέ πλέον ε, κυρώσεις. Η ε, αρχή ανταγωνισμού, η δική μας, έχει αποδείξει την αξία της, έχει, δημιου... έχει ε, κυρώσεις και σε περιπτώσεις καρτέλ και σε περιπτώσεις ε, όπου είχαν προσυμφωνηθεί τιμές ε, και έχουμε οδηγήσει και υποθέσεις στα ποινικά δικαστήρια. Έχει σημασία ότι αυτές όμως οι αποφάσεις μπορούν να εκτελεστούν μόνο ε, μετά την επικύρωσή τους από ένα ποινικό δικαστήριο. Ε, αυτό είναι το σύστημα στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει όμως ότι το βάρος της απόδειξης είναι περίπλοκο. Έχει Όμω και πλεονεκτήματα. Έχει πια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτό το σύστημα. Το, το, το γεγονός, για παράδειγμα, ότι οι δίκε γίνονται δημοσίω, δίνει τη δυνατότητα στου πολίτε να αντιλαμβάνονται ότι τα αδικήματα αυτά είναι ε, σοβαρά. Όμως η χρήση του ποινικού δικαίου δεν ε, ε, είναι πρόσφοροι σε άλλου τύπου υποθέσεις, όταν για παράδειγμα υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ παραγωγών και διανομέων ή άλλου τύπου καρτέλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις συχνά ζητείται από τους ενόρκους ή από τους δικαστές να, λάβουν, να, έχουν άποψη και να λαμβάνουν αποφάσεις για ζητήματα ιδιαίτερως πολύπλοκα. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πιο πρόσφαρο να χρησιμοποιείται κανείς ε, να χρησιμοποιούνται τα αστικά δικαστήρια. Ωστόσο, στην Ιρλανδία υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Τα αστικά δικαστήρια δεν μπορούν να επιβάλλουν ε, χρηματικά πρόστιμα. Ε, Επομένω, χρειάζεται ένα, η δυνατότητα επιβολή διοικητικών κυρώσεων και ταυτόχρονα ε, κάποιο είδου εντολή η οποία να σταματάει τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Εάν είχαμε τη δυνατότητα σε ορισμένε περιπτώσεις να μην επιδιώξουμε την επιβολή προστίμου, θα το είχαμε πράξει. πρέπει κανεί επίση να λαμβάνει υπόψη του ποιε θα είναι οι επιπτώσει μια απόφαση, όχι μόνο σε σχέση με μία συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και σε σχέση και με τι υπόλοιπε. Γιατί εάν σε μια υπόθεση, για παράδειγμα, επιδιώξουμε να επιβληθεί πρόστιμο και την γλιτώσει η εταιρεία, ίσω αυτό να οδηγήσει και σε άλλε εταιρείε του ιδίου κλάδου να υιοθετήσουν παρόμοιε πρακτικέ. πιστεύουμε, όπως και άλλες εθνικές αρχές ανταγωνισμού, ότι θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε όλων των ειδών της διαδικασίας, ποινικέ, αστικές, διοικητικές, γιατί η καθεμία από αυτές είναι πιο κατάλληλη για συγκεκριμένο τύπο υποθέσεις. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο ζήτημα του κατά πόσον υπάρχει μια τάση προς μεγαλύτερη συγκέντρωση κτλ. Εμείς πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αρχών Ανταγωνισμού έχει λειτουργήσει πολύ αποτελεσματικά, είναι πολύ χρήσιμο και για εμάς και για άλλες εθνικές αρχές. Μαθαίνουμε πράγματα, μοιραζόμαστε πληροφορίες και μεταξύ μας και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στοιχεία, πληροφορίες, ε, βέλτιστες πρακτικές, τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων. Μας έχει βοηθήσει λοιπόν. Ε, η δικιά μας αρχή έχει επίσης αρμοδιότητες στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή. Μακάρι να είχαμε ένα αντίστοιχο δίκτυο με αυτό που έχουμε στον τομέα του ανταγωνισμού για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και με τις άλλες αρχές της, ε, στην Ευρώπη που ασχολούνται με την προστασία του καταναλωτή. Κύριος Είμαστε ο επόμενο που είναι καθηγητή στο Κολέγιο της Ευρώπης και επίσης είναι αντιπρόεδρος στην ε, αρχή του, του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει εμπειρία 30 ετή και πλέον ο κύριο ε, Μάτζεν επίσης είναι και μέλος της ε, αρχής συναγωνισμού των νήσων της Μάχης. Πολλές φορές μερικοί προτιμούν να υπάρχει μια ε, νομοθεσία που να αφήνει πολλά περιθώρια συνεργασίας και σύγκλησης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η συνεργασία προκύπτει αβίαστα τότε που δεν επιβάλλεται. Δεν είναι εδώ να επιβληθεί η ευθυγράμμιση των ενδιαφερομένων. Αλλιώ η συνεργασία δεν είναι αυθεντική. Γι' αυτό σας λέω ότι να υπάρχει ε, ένα σχετικό ε, δίκτυο θα πρέπει να έχει δύο άξονες. Ανεξαρτησία και έγκαιρη ε, επισήμανση των διαφορετικότητων. Άρα, επομένω, δεν είναι πανάγια το να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. Οπότε ο στόχος μας είναι ECN, ακριβώς όπως τα αρχικά του δικτύου. Δηλαδή αποτελεσματικότητα, ανταγωνισμός και, ε, ε, και εφαρμογή του δικαίου. Πώς λέμε τα τρία ρο, στα αγγλικά reading, writing και arithmetic, αυτό είναι κάτι πολύ πιο βασικό βέβαια. Οπότε είναι βασικό ότι θα πρέπει να υπάρχει τέτοιου είδους αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου. Επομένως, τι είναι ακριβώς αυτή η μόνο επιθυντική θηρίδα που λένε για την ε, ε, επίοικια. Αυτό είναι ένα ευεργέτημα για τις εταιρείε που έχουν ε, παραβεί τον νόμο. Και έτσι να υπάρχει αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή του νόμου σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Έτσι όμως έχει κάποιο ατούτο το κράτος όσον αφορά με τα πολιτικά στοιχεία, είναι καλύτερη συνεργασία κατά την έρευνα Ήδη υπάρχει διαδικασία, ε, συνοπτική διαδικασία, όπου μπορεί να ζητηθεί από τις εταιρείε η ε, επίοικια. Χρειάζεται περισσότερη επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις πρώτες φάσεις της υποβολής αίτησης της επίοικιας. Οπότε, να, τι, ποια θα είναι που θέλουμε. Δηλαδή πάλι ECN στα ίδια αρχικά που σημαίνουν όμως ότι χρειάζεται έγκαιρη επικοινωνία. Για να δούμε τώρα τι είναι με τις κυρώσεις. Ε, είδαμε στη δική μας υπηρεσία ότι χρειάζεται μια αποτελεσματική και αλογική λειτουργία όσον αφορά την επιβολή προστήμων. Επίσης χρειάζονται κάποιο είδους δικονομικές εγγύησεις. Ακριβώς αυτό θα πρέπει να κάνει και το δίκτυο ανταγωνισμού. Ε, έχουμε ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων στην υπηρεσία μας και ε, έχουν προσβασιμότητα στη δικογραφία η διάδικοι, αλλά είπαμε ότι και πέραν των ε, προφορικών διαδικασιών, το πιο βασικό είναι η επικοινωνία. Υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση στις αποφάσεις και αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τις αποφάσεις μετά από διενέργεια συμβασμού, commitment decisions. Τι θέλουν. Πάλι εδώ πέρα το κλειδί είναι η επικοινωνία. Και οπότε πολλές φορές, έχουμε πολλούς περιορισμούς επί του ανταγωνισμού και ε, ε, τελικά η κάθε προσπάθεια καταλήγει σε μία από τα ίδια. Οπότε έχουμε πολλές πρακτικές που θα πρέπει να αναλυθούν ε, ανάλογα με το τι αρνητικά αποτελέσματα προκαλούν. Άρα θα πρέπει στο δίκαιο ανταγωνισμού να επικοινωνούμε όσο γίνεται σε πιο πρώιμη φάση, να καταλάβουμε τι ισχύει ε, σε κάθε υπόθεση, να συνεργαστούμε ούτω ώστε οι υποθέσεις να κρίνονται με έναν λογικό συνεπή τρόπο. Άρα χρειάζεται να έχουμε κάποιες μεθοδολογίες επιβολής προστήμων και θα πρέπει να έχουμε ένα κοινό ε, σώμα δικαίου όσον αφορά την βαρύτητα των ε, παραβάσεων. Επίση να αποφασίσουμε με νέο τρόπο τι γίνεται σε περίπτωση παραβίασης του δικαίου από κάποια θηγατρική και τι γίνεται με το πρόστιμο που επιβάλλεται στην ε, μητρική εταιρεία. Επίσης θα πρέπει να δούμε τα ελαφρυντικά ή τις επιβαρυντικές περιπτώσεις που συντρέχουν, οπότε θα πρέπει Να σκεφτούμε επίσης ότι οι διάδικοι πολλές φορές δίνουν πληροφορίες ε, γέρος ή καθυστερούν επίτηδες για να παρελκύσουν. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα, θα πρέπει να υπάρχει και ευελιξία που μας παρέχουν οι διαδικές στα αστικά δικαστήρια. Χρειάζεται νομοθετική λύση όταν δεν μπορούμε να έχουμε σύγκληση με εθνικές ρυθμίσεις. Πάλι εδώ είναι θέμα επικοινωνίας και κάθε μεταρρύθμιση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εθνική παράδοση και τις ε, εθνικές αρμοδιότητες. Να υπάρχει αναλογικότητα και να υπάρχει ε, συμφωνία όσον αφορά το μέγεθος, το εύρος και το βάθμισης εν κατακλείδη. Είπαμε ότι στην ε, Παλήρια, στην Άμποτη ε, σηκώνονται οι πέφτουν, χαμηλώνουν τα πλοία και εγώ θα προτιμούσα επομένω να το λάβουμε αυτό υπόψη και να έχουμε τα ελάχιστα πρότυπα. Άρα, να έχουμε ε, δυναμική στάση, έγκαιρη επικοινωνία και έτσι να πάμε προς το σκοπό μας που είναι η αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα ο τελευταίος να επιθυμίσω πριν δώσω το λόγο στον τελευταίο μιλητή ότι έχετε τις κάρτες σας για να πάρετε το λόγο. Παρακαλώ συμπληρώστε τις αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Οι περισσότεροι που έχουν ζητήσει το λόγο μέχρι στιγμής ε, είναι ευρωβουλευτές. Άρα θέλω να ενθαρρύνω τους άλλους συμμετέχοντες επίσης να παρέμβουν. Τελευταίος ομιλητής είναι ο Τζέρβιν Βαν είναι δικηγόρος ανταγωνισμού για 25 χρόνια. Είναι δικηγόρος στο γραφείο Link Latter στις Βρυξέλλες. ετέρος αυτό το δικηγορικό γραφείο και εκπροσωπεί ε, διάφορους ε, σε υποθέσεις ε, έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομες αγωγικές παρατηρήσεις για τα θέματα επίοικειας και τη σχέση μεταξύ των ευρωπαϊκών προγραμμάτων επίοικειας και των αντίστοιχων εθνικών. Θα αναφερθώ στα εξή σημεία. Πρώτον, όπως υπόθηκε, τα προγράμματα επίοικειας είναι σημαντική δυνατότητα στην εργαλειοθήκη εφαρμογής των ρυθμιστικών αρχών Άρα έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές να έχουν αποτελεσματικά προγράμματα ε, Αλλά για να είναι αποτελεσματικά πρέπει να είναι ελκυστικά για τους ενδεχόμενους αφορομένους. Να τους δίνουν κίνητρα για να συμμετάσχουν σε αυτά. Και το βασικό για αυτά, γι' αυτό για να είναι ελκυστικά, είναι η ε, προβληψιμότητα. Τι σημαίνει αυτό. Μια επιχείρηση θα πρέπει να είναι βεβαία ότι αν είναι η πρώτη που θα παραδεχθεί κάποιο πρόβλημα και αν πληρεί τα κριτήρια, τότε θα υπάρξει ασυλία και για την επιχείρηση και για τους εργαζόμενους της. Το δεύτερο είναι ότι η δομή για την εφαρμογή του νόμου με τις παράλληλες αρμοδιότητες των Εθνικών Αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργεί ε, προβλήματα με την ε, προβλεψιμότητα. Εάν μια επιχείρηση κάνει αίτηση επίοικιας ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή η αίτηση δεν της χορηγεί ε, προστασία σε εθνικό επίπεδο. Και μπορεί να είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς. Εάν παραδεχθεί μια παραβίαση τύπου καρτέλ, είναι δύσκολο να προβλέψει εάν θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό σε ευρωπαϊκό εθνικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο έχει διατυπώσει κατευθύνες γραμμές για να απευθυνθούν στο σωστό επίπεδο οι επιχειρήσεις, αλλά υπάρχει μια δυνατότητα ε, ελιγμών και άρα ένας βαθμός αβεβαιότητας. Και έχουμε παραδείγματα όπου ορισμένες υποθέσεις αρχικά ξεκίνησαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά τελικά αντιμετωπίστηκαν σε εθνικό επίπεδο από μία ή περισσότερες αρχές ανταγωνισμού εθνικές. Το δίκτυο έχει ένα πρότυπο πρόγραμμα επίοικειας ε, που έχει κάνει πολλά για να μειωθεί η αβεβαιότητα που, προκύπτουν, ε, η αβεβαιότητα που προκύπτει από αυτό το διεπίπεδο πρόγραμμα επίοικειας. Και ε, το πρότυπο αυτό είναι η συνοπτική αίτηση που προβλέπει αυτό το πρόγραμμα. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε ακόμη σημαντικές δυσχέρειες να αναφερθώ στις δύο πιο σημαντικές. Πρώτα απ' όλα, η προστασία των εργαζομένων, των φυσικών προσώπων. Εν μια εταιρεία κάνει αίτηση σε ενωσιακό επίπεδο για επίοικια και αν υπάρξει αντιμετώπιση σε ενωσιακό επίπεδο δεν υπάρχει πρόβλημα για τους ε, εργαζόμενους. Αλλά εάν ε, το αίτημα αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο υπάρχει ενδεχόμενο να διωχθούν ε, φυσικά πρόσωπα, γιατί στα κράτη-μέλη προβλέπονται κυρώσει και για φυσικά πρόσωπα. Άρα έχουμε εδώ το πρόβλημα. Πώς θα προστατεύσουμε μέσω της συνοπτικής ε, διαδικασίας τα άτομα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. γιατί η συνεργασία, η διάθεση των εργαζομένων στην επιχείρηση, των στελεχών της επιχείρησης να συνεργαστούν είναι ζωτική. Υπάρχουν διάφορα θέματα. Αν αυτή η προστασία αφορά τα στελέχη, υπό ποιε συνθήκε, άρα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ένα άλλο θέμα είναι ότι τα προγράμματα επίοικες βασίζονται στην προϋπόθεση ότι η επιχείρηση που κάνει αίτηση θα πρέπει να έχει σε εθνικό επίπεδο το ίδιο επίπεδο προστασίας με το ενωσιακό επίπεδο. Βέβαια, είναι θέμα ε, του, ε, της επιχείρησης να υποβάλει τα σωστά αιτήματα σε κάθε επίπεδο. Αλλά εάν τα υποβάλει τότε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ταυτόσιμο τρόπο. Δυστυχώς. Επειδή η συνοπτική διαδικασία έχει εφαρμοστεί, έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με διαφορετικό τρόπο, Υπάρχουν περιπτώσεις, όχι συχνές, όπου ναι μεν ε, υπήρχε προστασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά όταν μεταφέρθηκε σε εθνικό επίπεδο, η προστασία αυτή δεν ακολούθησε. Και άρα εξετέθησαν. Τελικά λοιπόν, είναι σημαντικό να υπάρξει περισσότερη συνέπεια, περισσότερη εναρμόνιση και θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επιδιώξουν περισσότερη και βαθύτερη εναρμόνιση. Μέχρι τώρα έχει γίνει με ήπια μέσα αυτή η εναρμόνιση. Έχει λειτουργήσει σε έναν βαθμό. Αλλά για να ολοκληρωθεί, να κόψουμε το νήμα, πρέπει να υπάρξουν και νομοθετικές πρωτοβουλίες. Είναι προς το συμφέρον όλων. Γιατί θα οδηγήσει σε περισσότερη προβλεψιμότητα και κατά συνέπεια σε πιο αποτελεσματικά προγράμματα επίοικεια παντού στην Ένωση και σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο και σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Έφτασε τι πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Θα περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις και τα σχόλια από τους συμμετέχοντες από το κρατήριο. Πρώτος ομιλητής, κύριο Τσάνη, ο ε, εισηγητής μας το, για το 2016 για ζητήματα ανταγωνισμού. Σας ευχαριστώ. Καλωσορίζω αυτήν την πρωτοβουλία και νομίζω ότι μας δίνει μια μοναδική ευκαιρία να συμφωνήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε βασικές αρχές για την πολιτική ανταγωνισμού και να τις εξοχρονίσουμε. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε συγκεκριμένες υποθέσεις, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που χρειάζεται και να αντιμετωπίσουμε ε, και πιο συγκεκριμένα στην Ουγγαρία. Πρώτα απ' όλα την περίπτωση ε, εξαγοράς από το δημόσιο μιας επιχείρησης στον τομέα των σιδηροδρόμων, της κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών. Ε, εννέα επιχειρήσεις είχαν δημιουργήσει ένα καρτέλ. Σε μία επιχείρηση δόθηκε πρόγραμμα επικίας. η οποία ετύχανε να είναι διοκτησίας του Υπουργού Εξωτερικών. Έχω άλλη μια υπόθεση από την Ουγγαρία που δείχνει πόσο χρειάζονται κανόνες ο, στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών είναι ένας τομέας ο οποίος ε, αναπτύχθηκε, συνέλεξε όλες τις άδειες η κυβέρνηση, τις απέσπασε μάλλον από τις εταιρείε όλες τις άδειες και τις έδωσε συνολικά πακέτο σε μια εταιρεία που όλος τυχαίω την είχε ένας φίλος του Πρωθυπουργού. Και επίσης τα ζητήματα των δημοσίων προμηθειών. Σε όλες τις περιπτώσεις πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθεί η διαφάνεια στο ευρωπαϊκό επίπεδο, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιθανώς και με χρήση οδηγιών ευρωπαϊκών. Και κατά την άποψή μου πρέπει να δημιουργηθεί και ένα νέο ε, ε, σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δίνεται η δυνατότητα σε αυτό το επίπεδο ευρωπαϊκό να υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος εάν χρειάζεται να μπορεί και να ανατρέψει αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο εθνικό επίπεδο. Σας ευχαριστούμε. Ο επόμενος ομιλητής, ο κ. Σφάμπ. Έχω πολλές ε, ερωτήσεις. Θα τις θέσω και όποιος από τους ομιλητές του πάνελ θέλει να απαντήσει, ας το κάνει. Η πρώτη ερώτηση είναι κάτι που τον ανέφερα και στους προηγούμενους ομιλητές, στο προηγούμενο πάνελ. Είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη εναρμόνιση και νέους κανόνες ε, οι οποίες θα απευθύνονται στα κράτη-μέλη, στις ε, αρχές των κρατών μελών. Αλλά η ερώτησή μου είναι η εξής, δεν θα έπρεπε αυτοί οι κοινοί κανόνες να απευθύνονται και να εφαρμόζονται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε τελικά όλοι να δεσμευόμαστε από τους ίδιους κανόνες και στον τομέα των προγραμμάτων επίοικης και των ποινών. Ε, η δεύτερη μου ερώτηση σχετίζεται με τις παρατηρήσεις του κ. Κέρβεν στο στις παρατηρήσεις που είχαν στο τέλος όσον αφορά τα κίνητρα. Υπήρξε για του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο πριν από δύο-τρία χρόνια ε, για μια οδηγία που σε άρθρο της έδινε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις εθελοντικά να αποζημιώσουν εκείνους που επλήγησαν από μια πρακτική τους. Εάν μια επιχείρηση όμως αποφασίσει να ακολουθήσει ένα τέτοιο θελοντικό πρόγραμμα επιζημίωσης. Δεν θα έπρεπε να υποφελείται και από ένα πρόγραμμα επιοίκειας και να προβλέπεται μείωση του προστίμου που τυχόν της επιβληθεί από την Κομισιόν είτε από την Εθνική Αρχή. Και επίσης, λέμε ότι θέλουμε να ενισχύσουμε τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ τους. Δεν θα έπρεπε να φροντίσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στις αρχές ανταγωνισμού της εθνικές να ε, υπερασπίζονται τις αποφάσεις τους ε, και εναντί των δικαστηρίων. με ενισχύοντα με αυτόν τον τρόπο και την ανεξαρτησία του. Να του βοηθήσουμε λοιπόν να πυροσβήσουν τι αποφάσει του στα δικαστήρια. Κυρία Γκουλάρ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ενότητε ερωτήσεων πρώτα απ' όλα για όλου εμά που ενδιαφέρονται για τον ανταγωνισμό ε, σε σχέση με τις ε, κυρώσεις που πρέπει να διέπονται από ενίο τρόπο επιβολής. Έχουμε επίσης και την Τραπεζική Ένωση που αφορά μόνο την ε, Ευρωζώνη και οπότε τι θα γίνει συγκεκριμένα τον ανταγωνισμό. Εσείς πώς το βλέπετε, πώς είναι δυνατόν να έχουμε ε, ενιαία αγορά για να καλύπτονται όλοι. Επίσης και κάτι άλλο που κάνει το λιματοπή Βρυξέλλας Σε περίπτωση Brexit, τι θα συμβεί, συμφωνείτε ότι θα πρέπει να είναι μέσα ή να είναι έξω από την Ένωση. Βέβαια θα πρέπει να συμβαστούμε την θέληση του λαού και θα πρέπει να μην φοβόμαστε την αλήθεια ότι δηλαδή η απόφαση και το, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα έχει συνέπειες και για τις χρηματαγορές και για τον ανταγωνισμό. Ο πρόεδρος η κυρία Μπερμέχο έχει τώρα το λόγο. Καλημέρα και ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτή όλη η προβληματική για την σχετική αποτελεσματικότητα των κυρώσεων για τη συμμετοχή σε καρτέλ ή για αποζημίωση εάν κανείς ομολογήσει την παράβασή του. Πολύ ενδιαφέρον, αλλά το θέμα είναι τι όρια έχει αυτή η υπόθεση και η αποτελεσματικότητα μέχρι που φτάνει η ανεξαρτησία πρώτα-πρώτα όσον αφορά τις κυρώσεις χωρίς κυρώσεις βαριές σε περίπτωση παραβίασης δεν υπάρχουν κίνητρα να σπάσει ένα ολιγοπόλιο και αν δίνουμε στους πληροφοριοδότες εκτεταμένη προστασία αυτό μπορεί να είναι αντιπαραγωγικό. Στην Ισπανία τα πρόστιμα είναι 10% του τζίρου. Στη νομολογία πολλές φορές έχουμε σημαντικές εκπτώσεις από τις αρχικά επιβληθήσεις ποινές. Και τελικά ούτε λογικά του τα έχουμε, ούτε αποτροπή. Εσείς θεωρείτε ότι αυτή η τάση είναι γενικευμένη. Πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Τώρα, έχουμε την, την συναρμόνιση. Έχουμε δει τι ισχύει στην Ευρώπη έχουμε δει περιπτώσεις και έρευνες ε, πρόσφατες για τις πολυεθνικές, αν τελικά δεν είναι φραγκοδίφραγκα αυτά που επιβλήθηκαν. Άρα μπορούμε να έχουμε τέτοια κατόφυλλα κυρώσεων που να μπορεί η κοινωνία να προστατευθεί από τις πολυεθνικές. Δεύτερη ερώτηση τώρα. Αυτή όλη η συζήτηση για τις κυρώσεις αναφέρεται σε κάποια αγορά αυθεντικά ανταγωνιστική. Όμως, η αλήθεια είναι ότι πολλά ολιγοπόλια γίνονται σε κάποιες αγορές που θα έπρεπε να είναι ρυθμισμένες και το κράτος προστατεύει τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών. Να, για παράδειγμα, οι διάφορες εταιρείε ηλεκτρισμού στην Ισπανία ξέρουν όλοι και το ερευνά και οι κομισιόν ότι ε, ωφελούνται αυτές οι, οι εταιρείε από τιμολογική πολιτική και επιβαρύνονται η, βιομηχανία και τα νοικοκυριά. Επίσης έχουμε την απόσβεση των παλαιών ε, υδροελεκτρικών ε, εγκαταστάσεων, έχουμε το πυρηνικό μορατόριο και γι' αυτό σας λέω, και αυτό έχει σχέση και με την πρώτη ομάδα ομιλητών δεν θα έπρεπε αυτοί που βάλουν τις κυρώσεις να λάβουν υπόψη σφαιρικά το τι γίνεται από πλευράς αρμοδιοτήτων ερευνητικών των αρχών ανταγωνισμού και να έχουν ε, επίσης αυτοί που παρέχουν ε, ε, υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος να διέπονται από διαφάνεια και κατά λίγο. Επίσης, η τιμολογική πολιτική και τα κέρδη των εταιριών θα πρέπει να είναι κριτήρια βασικά για να καταλήξουμε στο αν υπάρχει ολιγοπόλιο και να επιβάλλουμε τις σχετικές κυρώσεις. η ζητήσει το Κοινοβούλιο ε, να υπάρξει ε, πιο υγιής ανταγωνισμός και να υπάρχουν ε, παρατηρητές σε κάποιους τομείς όπως η γεωργία και να αποφύγουμε την στρέβλωση του ανταγωνισμού αλλά και διανομή. διανομής. Ε, ευχαριστούμε λοιπόν και τώρα από κάποια κρατικό φορέα. Κυρία Ορτή, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέγομαι Μαρία ορτή, είμαι από το Συμβούλιο και την Αρχή Ανταγωνισμού στην Ισπανία. Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για αυτή την πρωτοβουλία. Είναι μια πρωτοβουλία ιδιαίτερα σκόπιμη σε αυτή τη συγκυρία και ε, πολύ χρήσιμη. Από τότε που εγκρίθηκε ο κανονισμο 1 1-2003, σε αρχέ Ανταγωνισμού και Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργαζόμεθα πολύ στενά και το παρελθόν τη συνεργασίας των Εθνικών Αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια ιστορία επιτυχιών, πολύ θετικέ ανταλλαγέ πληροφοριών και επίσης ε, και η εφαρμογή των προγραμμάτων επίοικια είναι πολύ θετικές, έχει πολύ θετικέ επιπτώσει παρά του περιορισμού. Αν καταφέρουμε να αποφύγουμε αυτούς τους περιορισμούς, να καταλήξουμε σε κοινά στοιχεία, τότε η εργασία των εθνικών αρχών ανταγωνισμού θα είναι καλύτερη. Και αυτό θα ωφελήσει και την ασφαλεία δικαίου. Για τα προγράμματα επίοικειας θέλω να τονίσω πόσο σημαντική είναι η πολιτική κυρώσεων, ούτω ώστε τα προγράμματα αυτά να είναι πράγματι αποτελεσματικά. Και εδώ είναι βασική συνεργασία γιατί είναι το πιο σημαντικό μέσο που έχουν οι αρχές ανταγωνισμού έναντι των πιο επιβλαβών πρακτικών, των καρτέλ. Η πολιτική λοιπόν καθορισμού των κυρώσεων είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να υπάρξει σωστή ισορροπία μεταξύ αναλογικότητας και αποτροπής. Ήδη αναφέρθηκαν αυτά. Και αυτή η ισορροπία πρέπει να βασίζεται σε κοινέ προδιαγραφέ, ενωσιακέ κοινέ προδιαγραφέ, στα πλαίσια τη εσωτερική αγορά. Μόνο έτσι θα υπάρχουν ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού. Και μόνο έτσι τα προγράμματα επιοίκειας θα μπορέσουν να εφαρμοστούν και μόνο έτσι θα εφαρμοστεί σωστά και ισότιμα η πολιτική ανταγωνισμού παντού στην εσωτερική αγορά. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω τους ομιλητές αν μπορούν να μου πούν λίγο περισσότερα για το ποιες είναι αυτές οι ελάχιστες κοινέ προδιαγραφές για τα ανώτατα όρια των κυρώσεων και για τη μεθοδολογία υπολογισμού τους που να θεωρούν κατάλληλε ε, αρχές για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η πολιτική. Ευχαριστώ πολύ ο πρόεδρο. Brian Hayes. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ χαιρετίζω αυτή την πολύ σημαντική ακρόαση που έχουμε σήμερα. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν τον λόγο. Άκουσα την προηγούμενη συζήτηση από το γραφείο μου και άκουσα πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα θέλω να τονίσω η επιτυχία της Ευρώπης και η επιτυχία μικρών ανοιχτών οικονομιών όπως η δική μου, όπως είπε και ο δικός μας εκπρόσωπος, έχει ζωτική σημασία για την πολιτική ανταγωνισμού. Και η πραγματική ανάγκη είναι να διασφαλίσουμε ότι τα τοπικά συστήματα εφαρμογής λειτουργούν και να φαίνεται ότι, ότι λειτουργούν για να υπάρχει σωστός ανταγωνισμός σε αυτά τα κράτη-μέλη. Και το δεύτερο, η εργασία του δικτύου δημιουργεί νέες δυνατότητες, μας επιτρέπει να μάθουμε από την πύρα διαφόρων χωρών, διαφόρων αρχών, άνα κράτος μέλος, ζωτικής σημασίας. Και μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα ότι μελλοντικά θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ορισμένες υποθέσεις να τις εξετάζει η μία ή η άλλη αρχή για να μπορέσουμε να ε, ευθυγραμμίσουμε τις διαδικασίες. Να υπάρχει δηλαδή συνέπεια στις αποφάσεις. Για την Ιρλανδία και την Επιτροπή μας, η γι' αυτό, αναφέρθηκα ήδη στις κυρώσεις και με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι εκβάσεις κάποιων ε, πολύ ε, γνωστών υποθέσεων υψηλού επίπεδου. Είπε η αρμόδια ότι οι ποινές φυλάκισης ήταν με αναστολή σε όλες τις περιπτώσεις. Γιατί το λέω αυτό. Ορισμένε υποθέσεις έχουν ε, τεράστια απήχηση στην κοινή γνώμη. Πρέπει δηλαδή αυτές οι καταχρήσεις ε, δεσπόζουσας θέσεις, να αντιμετωπίζονται. Και η κακή συμπεριφορά μπορεί να αλλάξει μόνο μέσω κυρώσεων. Οπότε τίθεται το ερώτημα, είναι επαρκείς οι κυρώσει που έχουμε, είναι κατάλληλε, είναι οι σωστέ. Μήπω πρέπει ορισμένοι να μπουν μέσα για να σταλεί το σωστό μήνυμα. Είναι σημαντικό, πρέπει να το δούμε αυτό. Αλλά πέρα από αυτό, επίσης θέλω να τονίσω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα την εργασία της Ιρλανδικής Αρχής Ανταγωνισμού, αλλά και άλλων. Και τονίζω ότι πρέπει να συνεργαστούμε στενότερα, περισσότερο συντονισμό με όλους τους συναδέλφους παντού στην Ένωση, για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι δεσπόζουσες θέσεις κάποιων εταιριών καταγγέλλονται και καταδικάζονται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σουλάνακαν. Πολύ ενδιαφέρουσε οι παρουσιάσεις. Έχω μια, ε, ερώτηση για την κυρία Γκόγκενς. Είπατε ότι είναι πολύ σημαντική η πολιτική για τον ανταγωνισμό στην Ιρλανδία. Συμφωνώ πλήρω. Είπατε επίσης ότι η Ιρλανδία έχει αποδείξει ότι επιβάλλει αυστηρές ποινές και καταπολεμά τα καρτέλ. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Θα ήθελα να μου το εξηγήσετε καλύτερα. Αναφερθήκατε σε 33 υποθέσεις. Αλλά αυτές οι υποθέσεις αναφέρονται σε χρονιές όπως το 2006-2008, στην περίπτωση ε, μέχρι και ε, εταιρείε πετρελαιοειδών είχαν επιπρόστιμα 7.000-8.000 ε, ευρώ. 7.500 ευρώ πρόστιμο είναι δυνατόν να ήταν τόσο μικρό το κέρδος μιας εταιρείας πετρελαιοειδών που δημιούργησε καρτέλ στην υπόθεση της ε, εταιρείας Ήτρα. 20.000 ευρώ. Χωρίς, ε, και, και μάλιστα ανατράπηκε η ποινή το 2008. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσει κανεί καρτέλ στην Ιρλανδία για να έχει κέρδο 20.000. Επομένως, αν το, δει η επιχείρηση από πλευράς οικονομικής, μάλλον του συμφέρει να παραβιάζει την αντιμονοπολιακή νομοθεσία. Επομένως, πώς μας λέτε ότι καταπολέματε τα καρτέλ. Το 2011 ε, είχαμε μία υπόθεση. Ε, συχνά αναφερόμαστε σε αυτές τις 33 υποθέσεις, αλλά στην πραγματικότητα αυτά είναι προϊστορία. Η πρόταση της κυρίας Φερνάντες ήταν ιδιαίτερο ενδιαφέρουσα και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για αυτήν. Το λοκουστάν. Ε, ε δηλαδή, μα είπατε ότι η χρήση των αστικών δικαστηρίων, η προσφυγή στα αστικά δικαστήρια θα μπορούσε και αυτή να είναι πρόσφορη. Έχουμε όλο και περισσότερα παραδείγματα που να μας το δείχνουν. Ε, όσον αφορά τον συνάδελφο Χέις, θα ήθελα να του ζητήσω να διαβάσει την ομιλία του ε, συναδέλφου Χόγκαν το 2005 στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο, όταν ξεκαθάρισε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, ότι η κατάσταση ήδη ήταν τραγική, ήταν κομική ε, και, δεν έχει βελτιωθεί από τότε. Επομένως διαφωνώ μαζί σας όταν λέτε ότι στην Ιρλανδία καταπολεμάμε τα κατέλ. Ανέκδοτο είναι. Δεν, είναι μια τέτοια, δεν έχουν έτσι τα πράγματα στην Ιρλανδία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές να ρωτήσουν πως κάποιος άλλος από το κρατήριο θέλει να ε, παρέμβει. Είμαι μήπως τυχόν κάποιος από τους ομιλητές του πρώτου πάνελ θα ήθελε να μιλήσει τώρα. Όχι από ό,τι φαίνεται. Ας ξεκινήσουμε ε, τον γύρο των απαντήσεων με την κυρία Έντουαρτς. Σας ευχαριστώ. Έντουαρτσον. Κάποιες χώρες Εκείνε μάλλον οι χώρε οι οποίε χρησιμοποιούν το σύστημα με τις διοικητικέ κυρώσει είναι οι σκανδιναβικές, είναι οι μικρότερες ανοιχτέ οικονομίες και αυτό μου φαίνεται ενδιαφέρον. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στο ερώτημα του κ. Σουάμπ, αν ορθά το κατάλαβα. Ε, χρήσιμο θα ήταν οι διαδικασίε λήψη αποφάσεων να είναι εναρμονισμένε ή, εν πάση περιπτώσει, παρόμοιε. Αλλά το ερώτημα που τίθεται. Εάν το ερώτημα μάλλον που είναι αν θα πρέπει στις εθνικές αρχές να έχουμε ακριβώς τις ίδιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα. Δεν υπάρχει στη Σουηδία μια νομοθεσία η οποία οποία να μας εξαναγκάζει να συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ίσως είναι ένα ενδεχόμενο που πρέπει να εξετάσουμε. Από την παρέμβαση του κυρίου, της κυρίας Λόπες ε, κατάλαβα ότι πολλές φορές διαπιστώνεται ότι η ποινή είναι πολύ χαμηλή και θα θέλαμε γι' αυτό το λόγο να τις εναρμονίσουμε. Προσωπικά είμαι δικαστή και ξέρω ότι δεν είναι δυνατόν να εξαναγκάσουμε τα δικαστήρια σε διαφορετικέ χώρε να λαμβάνουν τι ίδιε αποφάσει. Είναι και ζήτημα αναλογικότητα, είναι και ζήτημα επικουρικότητα. Αυτά από την πλευρά μου. Ευχαριστώ. Κύριε σα ευχαριστώ. Θα σταθώ σε τρία σημεία από αυτά που ανέγυψαν. Συντονισμό, επίκαια και κυρώσει. Το είχα πει και στην ενσύχησή μου για τον συντονισμό. Αυτό που θα ήθελε ο επιχειρηματικό κόσμο να δει είναι το δίκτυο ανταγωνισμού να αποτελέσει την βάση για πιο καλό συντονισμό και πιο ε, συνεπή ε, προβληματική σε σχέση με τα μέσα της εξουσίας του των εθνικών αρχών. Να υπάρχει διάλογος δηλαδή μεταξύ εθνικών αρχών, του δικτύου, ε, οπότε ωφελούνται οι επιχειρήσεις και κυρίως όταν μιλούμε για τις ε, διαδικασίες της επίκης κλπ. Οπότε και έτσι να ξανοιχτεί κάπως αυτό το δίκτυο και προς επιχειρήσεις και προς καταναλωτές. Οπότε και να αποκτήσουν περισσότερη επαφή με την επιχειρηματική πραγματικότητα και άλλων χωρών οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού. Τώρα σε αυτό που ο κύριο ε, Σβάμπ ε, για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το είπα και αυτό στην αρχή, ότι θα πρέπει να είσαι κατευθυντήριας τις άρεστες πρακτικές. Αυτό είναι μια σωστή αφετηρία. Εάν αυτά τα εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιστρέφεται το ερώτημα. Για την επίκη τώρα. Εδώ πάντοτε είναι και θέμα ε, ηθικής και θα πρέπει να πούμε ότι κανένας δεν του αρέσει ε, να του επιβάλλουν κάτι, αλλά αν θέλει να είναι ρεαλιστής, τότε θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι με την επίοικια αποκαλύπτει, ξεμπροστιάζει κανείς τα καρτέλ. Και ε, αν φεσμοθετεί το, το αυτό μπορεί να είναι κίνητρο. Μπορεί, μπορεί αυτό να, να χορηγηθεί, να προβλέπει το καταδίκτυο για κάποιες εταιρείε. Τώρα, το κατά το σύστημα δίνει κίνητρα σε εταιρείε να βγαίνουν, να καταγγείλουν, να αποκαλύψουν, να ομολογήσουν. Ας είναι και μόνο μονοπευθυντική θηρίδα και σε περίπτωση καρτέλ. Να ξέρει μόνο ότι μια εταιρεία ότι αν πάει και προσφύγει σε κάποια αρχή ανταγωνισμού, σε οποιαδήποτε αρχή ανταγωνισμού, ότι μετά δεν θα διωχθεί. Τώρα όσον αφορά τις ε, κυρώσεις, τις ποινές, αν ε, το σύστημα των ποινών αρκεί, είναι αρκετά βαριές οι ποινές που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίση δημιουργούνται παντού αυτές οι ποινέ. Να επομένω τα αντικίνητρα και η αποτροπή. Δεν μπορώ να σχολιάσω το τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα πρέπει οι ποινέ να αρκετά βαριές που να αποτελούν αποτροπή. Αλλά εμεί θεωρούμε ότι η αποτροπή δεν επιτυχάνεται μόνο από το πόσο βαριά είναι μια ποινή. Είναι επίση και το θέμα του κατά πόσον κάποιο παραβάτη φοβάται ότι θα θα πιαστεί. Και βέβαια μπορεί και από ποινική διαδικασία να προκύψει χρηματική ποινή. Αλλά είναι το θέμα ε, βέβαια του πόσες υποθέσεις καταλήγουν σε ποινικό δικαστήριο. Αυτά για τις ε, κυρώσεις ποινές. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκόγκεν. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα υπόθεση και πολλοί εκφράστηκαν ε, υπέρ κάποιου βαθμού εναρμόνισης με ήπια ή μη μέσα. Φυσικά μέσω του δικτύου προσπαθούμε να επιτύχουμε πολύ ήπια εναρμόνιση, αλλά ορισμένα έχουν να κάνουν με τη φύση του δικαστικού συστήματος, όπου τα ήπια μέσα έχουν περιορισμένη επίπτωση. Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, επειδή το σύστημά μας είναι ποινικό ε, μέσω απαγγελία κατηγοριών δεν υπάρχουν ε, θέματα επίκαιες. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στους δικαστές να είναι επίοικοι. Αυτοί αποφασίζουν. Εμείς απλώς κάνουμε την προκαταρκτική έρευνα και μετά την αποστέλουμε στην εισαγγελία ο οποίο αποφασίζει για το αν θα ασκηθεί δίωξη. Και φυσικά κατόπιν ε, οι ένορικοι αποφασίζουν επί της ενοχής και οι δικαστές επί των ποινών. Ναι, είναι χαμηλά τα πρόστιμα, αλλά δεν το ελέγχουμε εμεί αυτό. Υπήρξαν και ποινέ φυλάκιση, αλλά όλε με αναστολή. Νομίζω ότι ένα πέρασε μια βραδιά στη φυλακή γιατί δεν πλήρωσε το δικαστήριο, άρα ήταν για λόγου. Ε, για λόγους μη συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι έχουμε μια ε, ολόκληρη γκάμα κυρώσεων ούτως ώστε ε, η ποινή να αντιστοιχεί στο έγκλημα. Ευχαριστώ κύριο Μάρσαν. Ευχαριστώ. Όταν ήμουν ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Office of Fair Trading της Υπηρεσίας για δίκαιο, ε, δίκαιες συναλλαγές πρέπει να πω ότι στην αρχή ήμουν επιφυλακτικός αλλά στην πράξη λειτουργεί καλά το σύστημα το είπαμε και προηγουμένως, οι εθνικές αρχές δεν θα έπρεπε να λειτουργούν, δεν λειτουργούν σε πολιτικό κενό. Οι διαδικασίες μας είναι απλώς δυνατότητα ε, επικοινωνίας και αλλοκατανόησης για να δούμε τι δεν λειτουργεί σωστά και μας βοηθάει να αποφύγουμε τη δημιουργία πολιτικής πίεσης. Δεν αφορά την επιλογή των αποφάσεων, συγγνώμη, των υποθέσεων και την ε, απόφαση. Βέβαια επιλέγουμε με ποιον θα ασχοληθούμε με βάση τα κριτήρια που έχουμε. Οπότε οι δυνατότητες που έχουμε για να ψάξουμε για παραβιά στην αγορά μας επιτρέπουν να βρούμε συγκεκριμένε λύσεις. Τι εναλλακτική λύση θα είχαμε. Ισχυρές πολιτικές παρεμβάσεις που δεν θα βασίζονταν ε, στα πραγματικά στοιχεία αυτό θέλω να το πω για τα θέματα διαφάνειας, γιατί είπα πολλά για την επικοινωνία προηγουμένως. Για τις συνοπτικές αιτήσει. είπα ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Οι νεότεροι ενημέρωση βέβαια θα ήταν καλή. Προτάσεις για το μέλλον λοιπόν. Θα ήταν σκοπιμότερο τα μέλη του δικτύου να συμφωνήσουν συγκεκριμένε προτάσεις για να βελτιωθεί η διαδικασία συνοπτικών αιτήσεων μέσω συνεργασία και διαλόγου. Και αν αυτέ οι προτάσει χρειαστεί να περάσουν από δημόσια διαβούλευση, βέβαια θα είχαμε πιο συγκεκριμένε απαντήσει επί συγκεκριμένων σημείων. Αντί να ασχοληθούμε με όλα τα θέματα των προγραμμάτων επί για τα πρόστιμα, ανώτατα όρια, ε, νόμιμα ή όχι. Σας είπα για, το, για την ευθύνη των ε, μητρικών εταιριών. Το σημαντικό είναι να δούμε και πού υπάρχουν ενώσεις επιχειρήσεων, ούτω ώστε να είναι όντως αποτρεπτικά τα πρόστιμα, εάν ε, οι παραβιάσεις έχουν γίνει από τις ενώσεις εταιριών. Και τα πρόστιμα πρέπει να λαμβάνουν πλήρως και τις πραγματικές συνθήκες ε, με τις οποίες διαπράχθηκε η παραβίαση. Τώρα τι ρόλο θα παίξει το Brexit, δεν θέλω να το αποφύγω. Είμαι πολίτη της Ένωσης, ε, συγγνώμη, πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν έχω βρετανική προφορά. Δεν ξέρω αν σα ενδιαφέρει λοιπόν η άποψή μου. Αλλά λόγω και της επίσημη θέσης μου δεν μπορώ να πάρω θέση. Αλλά σίγουρα θέλουμε να υπάρξει περισσότερη συνεργασία, πιο έγκαιρη ενημέρωση στα πλαίσια του δικτύου με όλου του ε, συναδέλφου μα. Παντού. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Τρία σχόλια, πολύ σύντομα. Τώρα έχουμε τον κύριο Σφάπ. το κατά πόσο στην οδηγία θα πρέπει να προβλέψουμε ότι όταν μια επιχείρηση εθελοντικά παρέχει αποζημιώσει, θα πρέπει να τη δίνεται ένα πρόγραμμα επιοικία. Κατά την άποψή μου αυτά τα δύο εργαλεία θα πρέπει να παραμείνουν ξεχωριστά. Είναι σημαντικό τα προγράμματα επιοικία να είναι ε, απλά, εύκολο να εφαρμοστούν, εύκολο να αποφασιστεί η εφαρμογή τους, ε, να μην εισάγουμε και νέους παρα, νέες παραμέτρους ε, που θα δυσχεράνουν τα πράγματα. Το δεύτερο, το ανέφερε και κάποιος ευρωβουλευτής, φαίνεται ότι κάποια πρόστιμα είναι πολύ χαμηλά Όσον αφορά όμω τις μειώσεις προστήμων που γίνονται προ επιχειρήσει, ο στόχο εδώ θα πρέπει να είναι να του δώσουμε κίνητρα και θα πρέπει να είναι ισχυρά τα κίνητρα αυτά. Ιδιαίτερα γνωρίζοντας ότι σήμερα στην Ευρώπη όταν διαπιστώνεται η ύπαρξη καρτέλ πολύ συχνά υπάρχουν και ατομικές αστικές προσφυγές Ε, επομένως αυτό είναι ένα σημαντικό βάρος για τις επιχειρήσεις που θα το καταγγείλουν. Και τρίτον, εάν χρειαζόμαστε περισσότερη εναρμόνιση ή ένα ενιαίο σύστημα για τα προγράμματα επίοικειας. Κατά την άποψή μου, είναι ότι κατά την άποψή μου λοιπόν, χρειάζονται κάποιες βασικές αρχές για τα προγράμματα επίοικειας οι οποίες βασικές αρχές θα πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο από όλους, με ένα αρμονισμένο τρόπο από όλους. Αυτό είναι η πρώτη προτεραιότητα, κατά την αποψή μου, να δημιουργηθεί ένα νομικό δεσμευτικό πλαίσιο για τα προγράμματα επίοικιας, το οποίο βεβαίως θα μπορούσε να, να, να τύχει και βελτιώσεων. Ανέφερα ένα παράδειγμα, να περιλαμβάνονται και τα φυσικά πρόσωπα στα προγράμματα επίοικιας θα μπορούσε αφού εισαχθεί ένα τέτοιο νομικά δεσμευτικό πλαίσιο η εναρμόνιση να ελέγχεται ε, κατά πόσο δηλαδή η εφαρμογή γίνεται με τον ίδιο τρόπο από όλους, να ελέγχεται και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, ο συνάδελφος έχει μια απάντηση, μάλλον κάποια σχόλια επιπλέον, κύριος Λομπράνο. Είπα στην αρχή, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Καταλαβαίνω ότι κάποιες από αυτές δεν αισθάνονται ότι χρειάζεται μεγαλύτερο συντονισμό. Το πρόβλημα όμω είναι ότι όταν δεν υπάρχει συντονισμός ή δεν δίνονται οι απατούμενοι πόροι στον συντονισμό, τότε οι επιχειρήσεις δεν βλέπουν ε, τις ευμενείς επιπτώσεις αυτού του συντονισμού. χρειάζεται μεγαλύτερη χρήση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού για να υπάρξει μεγαλύτερο συντονισμό των αρχών και όσον αφορά τα ζητήματα της όρθιης διαδικασίας. Και δεύτερον, για την σχέση μεταξύ προγραμμάτων επίοικειας και αποζημιώσεων. Ανέφερε ο κύριος Σφάμπ ότι προωθούνται συστήματα εναλλακτικά των δικαστηρίων για την επίλυση των αστικών διαφορών. Και επίσης τα στοιχεία που αφορούν στα προγράμματα επίοικειας πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικά. Αυτά είναι σημαντικά εργαλεία εάν θέλουμε να λειτουργεί το πρόγραμμα επίοικειας, αλλά επίσης θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το βασικό, η βασική διαδικασία ότι η επιχείρηση ζητάει να υπαχθεί σε ένα πρόγραμμα επίοικειας, μετά θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές και μετά θα έχει ασύλια. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Για να μπορεί ο διευθυντή μια επιχείρηση να παρουσιαστεί στο διοικητικό συμβουλίο τη επιχείρηση και να ε, πει ξεκάθαρα: Έχουμε δύο επιλογέ μπροστά μα, είτε να ε, ζητήσουμε το πρόγραμμα επίοικια, είτε όχι έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο και για το νομικό σύμβουλο τη επιχείρηση ποιε θα είναι οι επιπτώσει, να μπορεί να πει ξεκάθαρα στο διοικητικό συμβούλιο ναι ή όχι και να τι θα συμβεί. Να μην ξεκινήσει μια συζήτηση του τύπου ναι, ίσω εάν ε, ζητήσουμε το πρόγραμμα επιδίκεια από την Α ή Β Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού μπορεί να έχουμε διαφορετική ε, έκφαση τη υπόθεση. Ευχαριστώ. Πολύ χρήσιμη και η δεύτερη συζήτηση, ο δεύτερο γύρο. Τώρα να δώσω, τον κύριο στον κύριο... να δώσω τον λόγο στον κύριο Ιωάννη Λάτινμακερ για μερικέ καταληκτικέ παρατηρήσει. Ευχαριστώ την Επιτροπή σα, τον Πρόεδρο, τα μέλη και τη Γραμματεία που οργάνωσαν αυτή την ε, ακρόαση μαζί μας και σας ευχαριστώ όλους που είχαμε μια τόσο ζωηρή και επικοδομητική συζήτηση. Αυτό μας δίνει νέα ενάβσματα για την περαιτέρω εργασία μας. Είναι πολύ καλό που διαπιστώνουμε το Κοινοβούλιο, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού, αυτοί που ασχολούνται με αυτό το κλάδο, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία των πολιτών ασχολούνται ιδιαίτερα με την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές. και νομίζω ότι αν υπήρχε ανάγκη απόδειξης ότι οι εθνικές αρχές έχουν ε, βασικό ρόλο στο σύστημα η απόδειξη ε, είναι ενώπιον μας μετά τις συζητήσεις. Σίγουρα, στόχος μας είναι να λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά η εσωτερική αγορά προς όφελος και των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Όλα αυτά τα τονίσατε. Η εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές έχουν ευρύτερη επιλογή αγαθών και υπηρεσιών σε χαμηλότερες τιμές και διασφαλίζει ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ενιαία αγορά. Αυτό συμβάλλει στη δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθήκων για ανάπτυξη, απασχόληση και καινοτομία παντού στην Ένωση. Άρα πρέπει να βοηθήσουμε, να ενισχύσουμε την δράση των εθνικών αρχών, να τους χορηγήσουμε τα αναγκαία μέσα για τη σωστή λειτουργία τους. Όλα αυτά υπόθηκαν ιδιαίτερα εύγλωτα σήμερα το πρωί. Οι διακεκριμένοι ομιλητές μας, τους οποίους ε, θέλω και πάλι να ευχαριστήσω θερμά, έθεσαν πολύ σημαντικά θέματα και πολύ τόνισαν ότι χρειάζεται περαιτέρω δράση. Φυσικά δεν υπάρχει κανένα πρότυπο ενιαίας εφαρμογής. Πρέπει να τονίσουμε ότι χρειάζονται, χρειάζονται ευρωπαϊκές προδιαγραφές που να δίνουν περισσότερη δύναμη στη δράση των εθνικών αρχών. Επίσης τονίστηκε ότι η ανεξαρτησία είναι προϋπόθεση για πιο αποτελεσματικές ε, εθνικές αρχές ανταγωνισμού. Θα πρέπει να είναι σε θέση να παίρνουν αμερόλυτα τις αποφάσεις τους χωρίς καμία παρέμβαση είτε πίεση. Χρειάζονται λοιπόν διαφορετικές προϋποθέσεις ανεξαρτησίας οι οποίες περιγράφησαν. Χρειάζονται επιπλέον πόρους και αρμοδιότητες οι αρχές αυτές για να εντοπίσουν τις παραβιάσεις έγκαιρα και αποτελεσματικά. Έγιναν διάφορες ε, προτάσεις για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος ιδιαίτερα τα μέσα διερεύνησης που πρέπει να είναι ανάλογα με τις δυνατότητες απόκρυψης αποδεικτικών στοιχείων που έχουν οι επιχειρήσεις, κάτι που είναι ιδιαίτερη πρόκληση στην ψηφιακή εποχή. Ε, πολλά υπόθηκαν για κατάλληλε κυρώσει σε εθνικό επίπεδο. Χρειάζεται μια ευρία γκάμα κυρώσεων, όχι μόνο για παράδειγμα ποινικέ κυρώσει. Χρειάζονται και άλλου τύπου κυρώσει. Επιπλέον, τονίστηκε η σημασία των προγραμμάτων επί οίκειας. Γιατί μπορούν να μας βοηθήσουν να αποκαλύψουμε τα καρτέλ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα καρτέλ χρειάζονται ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότητα. Αν πρόκειται να ενθαρρυνθούν για να μας πλησιάσουν και να ομολογήσουν τις παραβιάσεις. Τονίστηκε ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο έκανε τα αναγκαία για να δοθεί περισσότερη νομική ασφάλεια. Αλλά χρειάζεται ακόμη περαιτέρω βελτίωση. Άλλα θέματα επίσης που τέθηκαν Ορισμένοι είπαν, για παράδειγμα, ότι η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και άλλων ρυθμιστικών αρχών, ιδιαίτερα προστασία καταναλωτών, πρέπει να ενισχυθεί. Και άλλοι είπαν ότι οι εθνικέ αρχέ ανταγωνισμού πρέπει να έχουν μεγαλύτερο ρόλο για τι κρατικέ βοήθειε. Όπω είπα είναι διαφορετικό το σύστημα, αλλά χρειάζεται να δημιουργήσουμε περισσότερο ισότιμε συνθήκε και οι εθνικέ αρχέ ανταγωνισμού μπορούν να παίξουν ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση. Κάτι ακόμη για την Τραπεζική Ένωση. Ο έλεγχο των συγχωνεύσεων, τα μέτρα αντιτράστ και τα μέτρα κατά το καρτέλ ισχύουν παντού. Και κρατικέ βοήθειε, όπου υπάρχουν ε, ειδικέ ρυθμίσει για τι ρυθμίσει τη ε, Τραπεζική Ένωση για την εξυγίανση των ε, τραπεζών. Έχει λάβει ο νομοθέτης λοιπόν τα αναγκαία μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις ανταγωνισμού στην ευρύτερη ενιαία αγορά. Τέλος, παραδέχομαι, όπως είπε και η Επίτροπος Βεστάγκερ, χρειάζεται περισσότερη χορήγηση σε εθνικό επίπεδο διαδικαστικών εγγύσεων. Αλλά να πω και κάτι ακόμη. Σε αυτούς που έθεσαν το θέμα του εάν και κατά πόσο η Κομισιόν πρέπει να θεωρήσει τους κανόνες της. Να κάνει μια αποτίμηση των κανόνων. Σας διαβεβαιώνω ότι ούτως ή άλλως πάντα έχουμε διαδικασίες συνεχής ε, αξιολόγησης. Από τότε που άρχισα να ασχολούμαι πριν από 15 χρόνια με τα θέματα αυτά, εκτός από τα άρθρα των συνθήκων, όλες οι άλλες ρυθμίσεις έχουν ε, επανειδωθεί μία, δύο και τρεις φορές. Άρα το γεγονό ότι σε αυτή τη φάση συζητάμε για το πώς ε, θα εξοπλίσουμε καλύτερα τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι η δική μας προσπάθεια για βέλτιστες πρακτικές και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες ε, έχει σταματήσει. Αλλά η βασική μας πρόκληση είναι πώς να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας σε εθνικό επίπεδο να έχουν τα αναγκαία μέσα που ήδη έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διάθεσή της. Οπότε, οπότε, Τι στοχεύουμε. Θέλουμε να κάνουν περισσότερα οι εθνικές αρχές. Θέλουμε να βελτιώσουμε το σύστημα ευρωπαϊκής εφαρμογής συνολικά. Νομίζω ότι οι συζητήσεις έδειξαν ότι αυτά τα δύο πρέπει να επιλεχθούν <coughs> εκ παραλίλου. Το σύστημα για να λειτουργήσει καλά πρέπει να λειτουργούν καλά όλα τα συστατικά μέρη του. Έλαβα υπόψη όλες τις απόψεις που ακούστηκαν σήμερα το πρωί και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μελετήσει προσεκτικά την περαιτέρω συμβολή ε, όλων μας πριν γίνουν περαιτέρω μέτρα. Με βάση αυτά που άκουσα από εσά και από άλλους ενδιαφερομένους, η Επίτροπος θα αποφασίσει τι περαιτέρω μέτρα είναι τα πλέον κατάλληλα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία ετοπίσαμε, όπως μας είπε σήμερα το πρωί. Υπάρχει δυνατότητα νομοθέτησης, αλλά πρέπει να έχουμε πιστικά πιστήρια από αυτού. Οπότε νομίζω ότι αυτά που ακούσαμε σήμερα το πρωί ήταν πολύ πολύτιμα. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους για τη συμβολή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που ε, μας καλέσατε να συμμετάσχουμε. Εμεί εμείς ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά, διότι και εγώ συμφωνώ ότι επρόκειτο για μια εκδήλωση πάρα πολύ σημαντική και να αξιολογήσουμε κατά πόσον συντρέχουν οι συνθήκες, οι προϋποθέσεις και αν χρειάζεται να προχωρήσουμε περαιτέρω ούτως ώστε να υπάρξει περισσότερη ποιότητα, περισσότερη αποτελεσματικότητα στο σύστημα επιβολής του δικαίου ανταγωνισμού και θα μπορούσε να πει κανεί ότι υπάρχει ευρεία συνένεση ότι έχουμε κάνει μικρά βήματα πρόοδου και αυτή η μερική έγκριση έχει αποδώσει, αλλά όμως θα πρέπει να έχουμε περισσότερη ομοιογένεια στην ε, εφαρμογή του δικαίου. Έχουμε επίσης και το θέμα της συνταγματικότητας του δικαίου ανταγωνισμού. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα αφενός όσον αφορά την ενιαία αγορά και αυτό φέρνει ομοιογένεια. Αλλά, απ' την άλλη μεριά υπάρχει αυτή η αποκέντρωση, αυτός ο συνδυασμός διαφορετικών εφαρμογών του δικαίου. Γιατί έχουμε κάποιες αποκλειστικές αρμοδιότητες όπως με την πολιτική μπορούμε να το συγκρίνουμε το προκείμενο ζήτημα. ή επίσης οι αποκλειστικές αρμοδιότητες προκύπτουν και από την Τραπεζική Ένωση. Άρα η βελτίωση και η αποτελεσματικότητα είναι κάτι το αναγκαίο. Και άρα προχωράμε τώρα σε μια τρίτη φάση μετά την προηγούμενη φάση της μερικής αποκέντρωσης και την πρώτη φάση της ε, κεντροκατηθενόμενης διαχείρισης. Τα είπε ξεκάθαρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει συνολικά να φροντίσουμε να υπάρχει λογική συνέπεια αναλογικότητα στο σύστημα λαμβανωμένων υπόψη βέβαια για τον ιδιωτυπιών του κάθε κράτους μέλους ποιότητα σημαίνει ομοιογένεια λύσεων έλεγε και ο Αριστοτέλης άρα θα πρέπει να δούμε όμως και τα αποτελέσματα αν δηλαδή έχουμε ομοιογένεια μέσων, για ποικιλία περιπτώσεων, κατά πόσον έχουμε ομοιογένεια αποτελεσμάτων. Όλα αυτά άρα τα λάβουμε υπόψη και να προχωρήσουμε έτσι σε διοικητική οργάνωση και να δοθεί και η διοικητική δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν στην πρόκληση. Υπάρχει βέβαια και ποικιλία απόψεων για το Ποιο θα ήταν, ο, ποιος ήταν η καλύτερη μέθοδος, περισσότερη αρμόνιση, περισσότερο συντονισμός. Νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο ο προβληματισμός μας. Το Κοινοβούλιο σίγουρα θα συνεργαστεί απολύτως μαζί σας. Να προστατευτούμε προς λύσεις που θα δώσει περισσότερη αποτελεσματικότητα στο δίκαιο ανταγωνισμού, να υπάρξει θεμητή οριονταγωνισμό και να υπάρξουν επίσης και τα κίνητρα για ανάπτυξη, για καινοτομία του πραγματικού συστήματος. Βέβαια, άλλο Ευαγγέλιο, η Τραπεζική Ένωση που και αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε μαζί σας. Έχουμε τώρα ένα όλος νέο νομοθετικό πλαίσιο αλλά επιβάλλεται αυτό το νομοθετικό πλαίσιο να είναι πολύ στεγανό. Και βεβαίως και θα τα πούμε και από αυτού μαζί. Αλλά να μην φεύγουμε από το σημερινό μας θέμα, διότι νομίζω ότι κάναμε ένα βήμα προς τα μπρος. Και το Κοινοβούλιο επιθυμεί την περαιτέρω εναρμόνιση και καινούργια μέσα εφαρμογής ε, του δικαίου από τις αρχές συνταγωνισμού. Πάρα πολύ σημαντική ήταν αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Και πάλι ευχαριστώ όλους όσους συμμετάσχουν. του ομιλητέ επίσης, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Ε, μια τεχνική λεπτομέρεια σύμφωνα με τα μέσα ασφαλεία τα οποία έχουμε οι εκπρόσωποι των αρχών ανταγωνισμού και οι άλλοι εξωτερικοί επισκέπτες για αυτή την ε, ακρόαση θα πρέπει όταν τελειώσει η συνεδρίαση να βγουν από την έξοδο του ισογείου αυτού του κτηρίου. Την έξοδο του ισογείου. Είναι καινούργιε ρυθμίσει, ε, καινούργιοι κανόνε ασφαλεία. Και πάλι σα ευχαριστώ. Πέρασε ακρόαση.